Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner vos places. Κυρίες και κύριοι, καθίστε. Παρακαλώ. Vous avez reçu... Έχετε ε, λάβει το σχέδιο ημερησίας διάταξης. Το newsletter, το δελτίο μας επίσης σας δίνει τις πληροφορίες για τις γλωσσικές διευκολύνσεις που είναι διαθέσιμες και έχετε επίσης στο φάκελό σας μια σειρά από έγγραφα υποδοχής που σας δίνουν τις ε, χρήσιμες πληροφορίες για τα νέα μέλη για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προϋπολογισμού και τα καθήκοντά μας. Έχετε επίση στη διάθεσή σας ένα απολογισμό της προηγούμενης θητείας του, της Επιτροπής Προϋπολογισμών που έχει προετοιμαστεί από τη γραμματεία μας, την οποία θέλω να ευχαριστήσω ως εκ τούτου. Το σχέδιο διορθωτικού για την ημέρησια διάταξη σας έχει διανεμηθεί στις 18 Ιουλίου. Πρόκειται για μια σειρά από τροποποιήσεις που έχουν κυρίως τεχνικό χαρακτήρα και εδώ υπήρξε συμφωνία με τα άλλα θεσμικά όργανα και υπήρξε στενή συνεργασία με την εισηγήτρια την κυρία Γκρέσλε. Βάσει του άρθρου 231 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το σχέδιο προτού ενδεχομένως το υποβάλει στην Ολομέλεια. Γι' αυτό το λόγο σας προτείνω αυτό το διορθωτικό να ε, παρουσιαστεί στην επόμενη Ολομέλεια, εάν δεν υπάρξει φυσικά αντίρρηση από κάποιο μέλος της Επιτροπής μας. Βλέπω λοιπόν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Το διορθωτικό λοιπόν αυτό αποτελεί αντικείμενο συνένεσης μεταξύ μας και γίνεται ομόφωνα δεκτό από όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Και ούτως εχόντων των πραγμάτων θα περάσουμε στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015 Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι το σημείο αυτό της σημερινής διάταξης συνδέεται με τα σημεία 4 και 5 για τα οποία δεν έχουμε διορίσει ακόμα εισηγητή για το μέσο ευελιξίας και για το Ταμείο Αλληλεγγύης συγκεκριμένα 4 και 5. Όπως ξέρετε το Συμβούλιο κατέληξε σε μια συμφωνία την προηγούμενη εβδομάδα σε επίπεδο Επιτροπής με Μονίμων αντιπροσώπων για να περικόψει κατά 2,1 δισεκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών και 100 εκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών το σχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί να σας εντυπωσιάσει ως πράξη του Συμβουλίου γιατί υπάρχει ήδη ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των δεσμεύσεων και των πληρωμών, των πιστώσεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών και βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει μια μείωση των πληρωμών κατά 2,1 δισεκατομμυρίων όταν οι πληρωμές περικόπτουν μόνο κατά 500 εκατομμύρια, συγγνώμη, όχι 100 εκατομμύρια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκουάρδεα Ζαβάλ, η οποία είναι η γενική συγγήτριά μας για το τμήμα 3 και μετά στην κυρία Χολμάιερ για τα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού. Κυρία Γενική Συγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να πω. Δεν έχω πολλά νέα για τον προπολογισμό 2015. Όπως πολύ καλά εξηγήσατε, το Συμβούλιο έχει ήδη υιοθετήσει μία θέση και αποφάσισε να κόψει τις πληρωμές και τις υποχρεώσεις, όπως ακριβώς είπατε. Και δεν είναι ότι μόνο δεν βάζει μέτρα για να λύσει το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με τις πληρωμές, αλλά αντίθετα κόβει τις πληρωμές για το 2015. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρόταση της Επιτροπής για τις πληρωμές ήταν το όριο, πραγματικά το όριο δυνατοτήτων που έχουμε από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε ότι θα ξεπεράσουμε σε περικοπές αυτό το όριο για το 2015. Πάντως, με τα ποσά που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο έκοψε τα ποσά αυτά, το 2,1 δηλαδή. Έτσι όπως βλέπουμε εμείς από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα πράγματα, θεωρούμε ότι το Συμβούλιο πρέπει επιτέλους να πάρει μια απόφαση λογική που να στέκει και να δεχτεί τους διορθωτικούς προπολογισμού που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λύσουμε έτσι σιγά σιγά το πρόβλημα των πληρωμών. Τώρα δεν έχουμε ενημερωμένα δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαντάζομαι το Σεπτέμβριο, θα μας παρουσιάσει την ακριβή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά τις ανάγκες του 2014 για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του 2015. Χθες στην Επιτροπή Πολιτισμού, που είμαι αναπληρωματικό μέλος, επίσης συζητούσαν το θέμα του προπολογισμού. Η υπεύθυνη εκεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λοιπόν, υπεύθυνοι για τον πολιτισμό, παιδί, αθλητισμό κτλ. προειδοποίησαν ότι αν δεν φροντίσουμε έγκαιρα να εγκρίνουμε του διορθωτικούς προπολογισμού, για άλλη μια φορά οι πληρωμές για το δεύτερο εξάμεινο του 2014 για τι υποτροφίε Έρασμο, για παράδειγμα, τίθενται σε κίνδυνο. Ελπίζω να μην ξαναβρεθούμε λοιπόν στην ίδια κατάσταση που είχαμε βρεθεί και πέρυσι, δηλαδή να μην έχουμε έγκαιρα λύσει και να αναγκαζόμαστε έτσι με έκτακτε συνεδριάσει να εγκρίνουμε διορθωτικούς προπολογισμού ε, στην ε, κόψη του ξηραφιού. Ελπίζω για τον έρασμο, αν μη τι άλλο, που είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα ευρωπαϊκής πολιτικής, να μην τεθούν σε κίνδυνο και πάλι. Ως εισηγήτρια και εμείς γενικά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχουμε μια ισχυρή τοποθέτηση όσον αφορά τις πληρωμές που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε. Βέβαια και οι υποχρεώσεις έχουν μεγάλη σημασία γιατί είναι οι πολιτικές που θέλουμε να αναλάβουμε. Οι υποχρεώσεις δείχνουν τις προτεραιότητές μας και οι πληρωμές δεν πρέπει να είναι απλώς και μόνο ένα τεχνικό στοιχείο, αλλά παρόλα αυτά οι υποχρεώσεις είναι αυτές που δηλώνουν ποιε είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε. Δυστυχώς, μέρος των προσπαθειών μας πρέπει να είναι η πειθό απέναντι στο Συμβούλιο για να μπορέσουν να πληρωθούν τα προγράμματα για τα οποία έχουμε αναλάβει δεσμεύσει. Οι πολιτικέ προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι σαφέστατε. Όπω είπαμε το Μάρτιο στι γενικέ κατευθυντήριε γραμμέ, πρέπει τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα να έχουν στη διάθεσή τους όσο γίνεται περισσότερα χρήματα, ώστε να μπορούν να γίνουν οι πληρωμές. Να μην περιμένουμε όπως έγινε παλιότερα, περιμένουμε από το 2008-2009 χρόνια μετά για να πληρωθούν. Είναι αυτό μεγάλο πρόβλημα για τα προγράμματα. Και αυτό βάζει και την Ευρώπη σε δύσκολη θέση, η οποία αντίθετα πρέπει να εξυγχρονίζεται, πρέπει να είναι σε θέση να ανταγωνίζεται τον υπόλοιπο κόσμο και όχι να έχει χαμηλότερους μισθούς και χαμηλότερα προσόντα. Αντίθετα, από πλευρά ευρωπαϊκού προπολογισμού λοιπόν πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να το καταφέρουμε αυτό, να βοηθηθούν οι χώρες μέλη και να φροντίσουμε τα διάφορα προγράμματα που θέλουμε, εκπαιδευτικά και άλλα, να προωθηθούν, ώστε η Ευρώπη πραγματικά να αποτελεί σημείο αναφοράς ή τέλος πάντων να ξαναείνει σημείο αναφοράς ανά τον κόσμο. 50% λοιπόν των προσπαθειών για τις υποχρεώσεις και 5% για τις ε, πληρωμές. Γιατί αν αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις αλλά μετά δεν μπορούμε να πληρώσουμε, καταλαβαίνετε ότι πάει στράφη η δουλειά μας. Και ένα μικρό σχόλιο, ακόμα κάποια στοιχεία να σας δώσω για ε, πειραματικά προγράμματα. Αποτελούν κάτι που αρέσει πάρα πολύ στους ευρωβουλευτές. Τώρα έχει περάσει η δεύτερη προθεσμία για την υποβολή προγραμμάτων. Ανάμεσα στους δύο γύρους λοιπόν, οι ευρωβουλευτές υπέβαλαν 117 τέτοια πειραματικά προγράμματα και 34 προπαρασκευαστικές δράσεις. 27, 24 νόμοι υπήρχαν είχαν ήδη, αλλά είναι καινούρια. 1.400.000 ευρώ. Έχουμε ήδη την πρώτη αξιολόγηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά. Ξέρετε ότι στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις που έχουν γίνει, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή τεχνικά να αξιολογήσει αν πρόκειται για κάτι που μπορεί να προχωρήσει ή όχι. Την έχουμε λοιπόν αυτήν την αξιολόγηση. Στον πρώτο γύρο βέβαια είχαν μείνει τέσσερις χωρίς αξιολόγηση. Το Σεπτέμβριο φαντάζομαι θα πάρουμε την αξιολόγηση αυτών των τεσσάρων που δεν αξιολογήθηκαν αρχικά, συν τη δεύτερη αξιολόγηση των υπολείπων. Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να ξέρετε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει ότι υπάρχει μια πολιτική προτεραιότητα να προχωρήσουμε με ένα από αυτά τα πειραματικά προγράμματα, Ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική η αξιολόγηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί μπορούμε να δώσουμε το πράσινο φω και να το πούμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προχωρήσει. Μία απαραίτητη προπόθεση είναι η αξιολόγηση, αλλά σα είπα ότι δεν φτάνει για να προχωρήσει όχι ένα πρόγραμμα. Πάνω απ' όλα σημασία έχουν, πιστεύω εγώ, οι δικέ μα πολιτικέ προτεραιότητε. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γενική Εισηγήτρια, για τις παρατηρήσεις σας. Νομίζω πως όντως ε, βρισκόμαστε στην αρχή της θητείας και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο επίπεδο των πληρωμών σε σχέση με τις υποχρεώσεις, διότι υποχρεώσεις που δεν ε, χρηματοδοτούνται μπορεί να φανούν ως απάτη. Και δεν μπορούμε να ανεχθούμε ότι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν υπάρχουν χρέη δεν προβαίνουμε στην εξόφληση των ε, ε τιμολογίων που πρέπει να πληρωθούν. 100 δις το 2010 και 134 το 2013 και η τάση είναι ανησυχητική. Ο κύριος Μάνκα θέλει το λόγο. Eh, Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που συνόψισε τα θέματα και να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί της ότι το βασικό και κυριότερο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δεσμευόμαστε, αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις και μετά δεν γίνονται οι πληρωμές για ε, ε, αρκετά χρόνια τέλεσα δήμαρχος ε, μιας πόλης και ξέρω τι θα πει όταν καθυστερούν οι πληρωμές. Εμείς κατασκευάζαμε σύνδεση ε, ανάμεσα σε δύο κράτη, γιατί σε δύο μάλλον ε, περιφέρειες, ε, γέφυρες προσπαθούσαμε να φτιάξουμε. Το 50% προερχόταν από τις δικούς μας πόρους και το υπόλοιπο το περιμέναμε. Αυτό ήταν τεράστιο πρόβλημα. Πριν από λίγα χρόνια πέρασε μια οδηγία όπου το Συμβούλιο ανέλαβε ότι θα καταβάλει τις πληρωμές εντός 10 ημέρου. Μετά αυτό έγινε 60 μέρες και τώρα το Συμβούλιο παραβαίνει το λόγο του. Τεράστιο πρόβλημα. Εάν δεν πληρωθούν στην ώρα τους τα έργα, τότε και οι Δήμοι δεν θα πάρουν τα λεφτά τους στην ώρα τους και πάει λέγοντας. Το 4% μόνο των επιχειρήσεων έχουν αρκετού πόρου στη διάθεσή του για να τα πληρώσουν όλα μόνα του και έχουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα διαρθωτικό και το Συμβούλιο αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσει ε, και το, το, την επίλυση αυτού του προβλήματος, το οποίο επανέρχεται ε, κάθε χρόνο. Η μόνη λύση που εγώ μπορώ να σκεφτώ είναι να εφαρμόσουμε τη δέσμευσή μας, να εφαρμόσουμε το σύστημα των ιδίων πόρων και ξέρω ότι ο κύριος Γιούνκερ ε, ανέλαβε να ολοκληρώσει το θέμα του φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριο Στόβαλτ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια Μία από τις πρώτες προτάσεις στην εισήγησή της ήταν αν το Συμβούλιο λάβει μια λογική απόφαση. Ακόμα και αν προέρχομαι από τη χώρα του Αϊβασίλη και θα έπρεπε να πιστεύω στα όνειρα και στους μύθους, δεν πιστεύω στη δυνατότητα τώρα το Συμβούλιο ε, εδώ κοντά να λάβει τέτοια λογική απόφαση. Για να δούμε ότι θα πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα, αν θα γίνει το θαύμα των Χριστουγέννων. Έχω να πω τα εξή για αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι κάποιε από τι υποχρεώσει που αναλαμβάνουμε είναι κάπω ε, τυχοδιοκτικέ. Γιατί ε, αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται συντόμως να υλοποιηθούν. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε πιο επιφυλακτικοί σε αυτό το τομέα. Γιατί αν ξεκολουθήσουμε να δείχνουμε πως είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο και πώς θα πανούμε τα χρήματα που δεν έχουμε, τότε το τέλος θα είναι πολύ λυπηρό. Όταν λέω ότι πρέπει να εξετάσουμε τις υποχρεώσεις, εγώ θέλω να ακούσω μία υποχρέωση από το Συμβούλιο και αυτό είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση. Γιατί αν ε, είναι κάτι το τελείως τυπικό, τότε θα είμαστε σε άσχημη θέση. Θα φαινόμαστε σαν ηλίθιοι εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και δεν θα ήθελα αυτό να συμβεί. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με αυτό το δύσκολο προπολογισμό του 2015 ε, βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο phasing in των νέων ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Μόνο το 20% των κονδυλίων θα δοθούν για τα νέα προγράμματα και το 40% για την ολοκλήρωση των παλιών προγραμμάτων. Και για να μπορέσουμε αυτό να το διαχειριστούμε, Δεδομένων των όσων γνωρίζω για την αυξανόμενη καθυστέρηση από το 2014, το κλειδί για την επιτυχή διαχείριση του 2015 είναι να έχουμε να γίνουν ε, ε, προσθήκες για το 2014 για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το κενό. Έπειτα θα έπρεπε να εστιάσουμε στις υποχρεώσεις και μετά να έρθουμε με τις πληρωμές για να μειώσουμε τις καθυστερήσεις. Το ανώτατο όριο για το 2015 είναι χαμηλότερο κατά 2 δις από ότι το 2014. Ε, και αυτό είναι πάλι δύσκολο γιατί η οροφή τώρα είναι 8 δις χαμηλότερα από ό,τι δαπανήθηκε από το περασμένο έτος. Βλέπουμε λοιπόν τις δυσκολίες και δεν βλέπουμε λύσεις για το 2014. Είναι αδύνατη αποστολή, είναι mission impossible να, να διαχειριστούμε σωστά το προπολογισμό. Έπειτα, οι περικοπέ τι οποίε έχει προβεί το Συμβούλιο είναι απόλυτα αντιφατικέ με τι δικέ του δηλώσει. Μπορώ να σα παραθέσω επιλεκτικά από το Συμβούλιο τον Ιούνιο για το τι έγινε δεκτό ήταν η στρατηγική ατζέντα για την Ένωση σε καιρού ε, αλλαγών και ότι θα πρέπει λέει, να επενδύσουμε στην οικονομία της ενέργειας ε, στο, για το μέλλον, να κινητοποιήσουμε και ιδιωτικό και δημόσιο χρήμα, να διευκολύνουμε τις, ξένε τις ξένες επενδύσεις κτλ. κτλ. Οι περικοπές είναι απόλυτη, σε απόλυτη αντίθεση με τα όσα δέχτηκαν οι κυβερνήσεις τον Ιούνιο 26 και 27. Αλλά η επιτυχής διαχείριση στην ουσία έγκυται στις προσθήκες που θα γίνουν για να γεφυρωθεί το κενό το 2014. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ. <clears throat> Κύριε Ζάνη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εισήγησή της. Εγώ είμαι ναι, αφιχθεί εδώ, στην κοινοβούλιο και στην Επιτροπή αυτή. Και όταν ε, μπήκα στην ουσία του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού πρέπει να σας πω ότι σοκαρίστηκα από το πρόβλημα των πληρωμών. Είναι ένα πρόβλημα ε, ψάχνοντας ανάμεσα στα κείμενα, ξεψηρίζοντάς τις, ε, ανατρέχει στο 2002. 12 χρόνια τώρα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, διονύζουν αυτό το πρόβλημα. Αν τα θεσμικά μας όργανα θέλουν να είναι αξιόπιστα, απέναντι στους πολίτες πρέπει να τηρούν τις υποσχέσεις τις οποίες έχουν αναλάβει και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Κατά τη γνώμη μου, η θέση του Συμβουλίου για τις προϋπολογισμό και τις πληρωμές για το 2015 είναι απαράδεκτη. Πρέπει να δουλέψουμε για να μειώσουμε αυτή την καθυστέρηση τους ώστε να καταστούν τα όργανα αξιόπιστα. Όπως έλεγε πριν και, το ο συνάδελφος, δεν είναι μόνο θέμα αξιοπιστίας, αλλά είναι και θέμα οικονομικό. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πληρώνει όσους έχουν ε, κάνει παροχή των υπηρεσιών, δεν πληρώνει τις υπηρεσίες και τους ε, τοπικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις και αυτοί δεν μπορούν να επενδύσουν, δεν μπορούν να πληρώσουν μισθούς και πέφτει σε ύφεση η οικονομία. Είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν είναι βιώσιμος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ξέρετε, η συζήτηση ξεκίνησε αμέσως μετά την παρουσίαση της ε, κυρίας Γενικής Υγήτριας και θέλω να δώσω και το λόγο στην κυρία Χολμάιερ, η οποία είχε ένα κόλλημα που την εμπόδισε να είναι παρούσα στην αρχή της συζήτησης. Αν θέλετε λοιπόν, μπορούμε να διακόψουμε μια στιγμή τη συζήτηση και να δώσουμε την ευκαιρία στην κυρία Χόλμαερ να συμπληρώσει τα λεγόμενα της εισηγήτριας, της κυρίας Γουαρδίας Ζαμπάτ και μπορούμε να συνεχίσουμε μετά. Εγώ θα πρέπει να σας μιλήσω για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρξαν διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε μια ειδική κατάσταση ίσως μέχρι το τέλος του έτους, γιατί είναι πολλά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία έχουν αποχωρήσει στις εκλογές του 2014 πάνω από τον μέσον όρο και όλα αυτά θα έχουν φυσικά και επιπτώσεις για το 2015 γιατί θα πάρουν κάποιες αποζημιώσεις μετάβασης τα μέλη αυτά τα οποία αποχωρούν ενώ συγχρόνως έρχονται τα νέα μέτρα και επίσης έχουμε ως μέρους συναδέλφους οι οποίοι έχουν, είχαν αναλάβει τον προϋπολογισμό και έχουν έχουν αποχωρήσει. Έχουμε μια προσαρμογή στο 1,8% και 0,4% πρόσθετα κονδύλια τα οποία θα χρειαστούν. Αυτά είναι περισσότερα από ό,τι είχαν προβλεφθεί στο παρελθόν. Πρέπει επίσης να συζητήσουμε για το κόστος των κτίριων, κατά πόσο θα τα αναβάλουμε για το μέλλον ή θα, αν θα υπάρξει μία ε, πληρωμή τους και εδώ στο οργανόγραμμα υπάρχουν 67 ε, θέσεις οι οποίες στη διοίκηση οι οποίες ε, διαγράφονται και επίσης έχουμε και το νέο στοιχείο ότι υπάρχει μια συμφωνία με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή οπότε υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και στους δύο προϋπολογισμούς και του Κοινοβουλίου και της ε, Επιτροπή των Περιφερειών. <clears throat> θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν να διευκριστεί καλύτερα ποιε θα είναι οι τελικές αλλαγέ στους προϋπολογισμούς των ε, δύο οργάνων αυτών, της ε, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπή των Περιφερειών, γιατί και τα δύο αυτά όργανα θα μεταφέρουν ένα τμήμα του προσωπικού στο Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται λοιπόν για αύξηση του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόκειται για μεταφορά θέσεων από το οργανόγραμμα αυτών των οργάνων στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Επομένως είναι σαν να παίρνει ένα πρόσθετο ποσό προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμεί, μέχρι τον ε, Σεπτέμβριο ελπίζουμε θα έχουμε τα τελικά ε, στοιχεία για τον αριθμό των μελών του προσωπικού που θα έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε και στους άλλους τέσσερις τομείς κάποια προβλήματα. Έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην, Επιτροπή, στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, από, όπου κατά την ε, απόψή μου το Συμβούλιο έχει επιφέρει δυσανάλογες και όχι απλώς οριζόντιες περικοπές και αυτό τη στιγμή που υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες δεν έχουν μπορέσει να καλυφθούν με στελέχωση νέου προσωπικού. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν και εκεί να δούμε ποια είναι η τελική <clears throat> κατάσταση ε, γιατί προς το παρόν υπάρχουν και θέσεις σε πρεσβείες και προξενία που δεν μπορούν να σε τις της ε, υπηρεσίε εξωτερική δράση που δεν έχουν καλυφθεί. Επίση, είχαμε συζητήσει μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου. Το Συμβούλιο είναι σαν να μην έχει διαβάσει τη δική του θέση για όλα αυτά και έχει περικόψει τα ποσά τα οποία είχε εγκρίνει προηγουμένω για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και εντωμεταξύ έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των υποθέσεων που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό σημαίνει ότι έχουν αρχίσει να καθυστερούν οι εκδικάσεις μέχρι τρία χρόνια πια. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι πρέπει να πληρώσουν πρόστιμα ε, της τάξεως ε, ευρώ και αν καθυστερεί η δίκη τρία χρόνια θα πρέπει το ποσό αυτό να αποδοθεί αν κερδίσουν τη δίκη με τόκους. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σοβαρά προβλήματα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα πρέπει να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά με το Συμβούλιο, γιατί το Συμβούλιο έχει απο... απομακρυνθεί από τη δική του αρχική θέση και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και κατά τα άλλα για τα άλλα τμήματα, για τις άλλες πτυχές του προπολογισμού υπάρχουν μικρά προβλήματα τα οποία μπορούμε αν χρειαστεί να τα συζητήσουμε και αυτά. Ευχαριστούμε κυρία Ολμάερ. Έχουμε μπροστά μας ένα άθλο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξάλλου και αυτό θα πρέπει να παίξει πλήρως το ρόλο του στα θέματα αυτά. Ο κύριος Ντάτσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα και εγώ η ίδια να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και να συγχαρώ φυσικά την, ε, τις εισηγήτριες που έχουν κάνει μια πολύ καλή εργασία για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα τώρα να συνοψίσω τη θέση μου σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα, ναι, θα ήθελα να υποστηρίξω την εξή άποψη ότι για τον προπολογισμό του 2015 αυτό το οποίο έχει αποφασίσει το Συμβούλιο είναι απόλυτα απαράδεκτο. Είναι απόλυτα απαράδεκτο γιατί το Συμβούλιο δεν βοηθάει καθόλου την επίτευξη λύσεων στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λεβαντόφσκι, αλλά ήδη σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων υποχρεώσεων. Αυξάνει συνέχεια το χάσμα αυτό, θέτει σε κίνδυνο κοινέ πολιτικές όπως είναι η πολιτική συνοχής και η αγροτική πολιτική και η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο δεν θέλει να δώσει καμία λύση, απλώς οξύνει περισσότερο τα προβλήματα αυτά. Επίσης θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα προβλήματα τα οποία αναδύονται στον προϋπολογισμό του 2015 δεν έχουν αντιμετωπιστεί. υπήρξε ένα συνολικό πλαίσιο για, τα για την πολυετή δημοσιονομική χάραξη προτεραιοτήτων, αλλά αυτή δεν ήταν μια θετική συμβιβαστική λύση που επετέφθη σε σχέση με τις πολιτικές προοπτικές, πολιτικές είναι μια πολύ μέτρια ε, συμφωνία. Και το Συμβούλιο μπορεί να είναι ένα από τα βασικά όργανα του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να λάβει υπόψη του Κοινοβουλίου, το οποίο βρίσκεται μόνο μερικές μέρες μετά από τις εκλογές και δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί πλήρως. Όλοι θέλουν περισσότερη Ευρώπη. Αυτό ζητήσαμε όλοι, αλλά το Συμβούλιο όταν πρέπει να δώσει περισσότερη Ευρώπη, το λέει φραστικά μεν, αλλά σε επίπεδο συγκεκριμένο, σε επίπεδο απτό, όταν πρόκειται για χρηματοδότηση, όταν πρόκειται για προπολογισμό, το Συμβούλιο θέλει ουσιαστικά λιγότερη Ευρώπη. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Γι' αυτό τον λόγο θέλω και πάλι να επιστήσω την προσοχή όλων στο ότι το Συμβούλιο και η Προεδρία του Συμβουλίου θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ουσιαστικά θέματα. Εκεί θα πρέπει να καταδείξει το Συμβούλιο ότι πράγματι υποστηρίζει περισσότερη Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο να δείξουν αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ επειδή ήδη ακούστηκαν πολλά, θέλω να περιορίσω τα σχόλιά μου στο γενικό προπολογισμό. Ευχαριστώ την για το σχόλιά τη. Οι υποχρεώσει ήταν ανέκαθεν πολύ σημαντικέ για την Επιτροπή Προπολογισμού, γιατί στην ουσία πρόκειται για δεσμεύσει για το μέλλον. Αλλά βέβαια, όταν συζητάμε το προπολογισμό του 2015, το πραγματικό πρόβλημα θα είναι πάλι το επίπεδο των πληρωμών. Και ήδη ακούσαμε πως το Συμβούλιο πιθανότατα θα θελήσει να περικόψει το σχέδιο προπολογισμού που προτείνει η Κομισιόν κατά περίπου 2 δις ευρώ. Πράγμα το οποίο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, ιδιαίτερα να αναγνωρίσουμε ότι ήδη μας λείπουν χρήματα, ότι ήδη οι περικοπές που προτείνονται θα, θα προσθεθούν ε, στην 1α και στη 4 που είναι προτεραιότητες για την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θα υπάρξουν λοιπόν σοβαρές επιπτώσεις. Τώρα, Δυστυχώ κάποια κάτι μέλη θα το αρνηθούν αυτό. Θα πούνε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και γι' αυτό είναι χρήσιμο για την Επιτροπή μα να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε του τομεί όπου βλέπουμε αυτά τα προβλήματα και να μα πει η Κομισιόν που πιθανώ θα υπάρξουν καθυστερήσει, που δεν θα γίνουν μάλλον πληρωμέ. Ήδη ακούσαμε ότι, για παράδειγμα, θα έχουμε ε, πρόβλημα με το έρασμο. Είτε σήμερα είτε σε κάποια μελλοντικέ συνεδρία θα πρέπει να δοθούν αυτέ οι λεπτομέρειε, ίσω και γραπτό, ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε στην Επιτροπή μα αλλά και στο Συμβούλιο, αλλά και στον κόσμο που εκπροσωπούμε, ότι αν δεν γίνονται οι πληρωμέ θα υπάρξουν ε, σοβαρές, σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσει. Σας ευχαριστώ. Έχουμε συζήτηση για το θέμα, είχαμε μάλλον την περασμένη Τετάρτη. Ήδη εκεί ε, ακούσαμε και αρχίσαμε να λέμε για το τι σκοπεύουμε να σεβαστούμε. Ο κύριος Δελανό, ευχαριστώ. Και εγώ, Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συγκήτρια που τόνισε τα σημαντικά θέματα και μας έδωσε ε, λαβή για προγραμματισμό. Εγώ πιστεύω, για τα... πιστεύω ότι το θέμα του προπολογισμού καθορίζει το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως καθορίζει την αναγνώριση από πλευρά των κρατών των πολιτών της ίδιας της Ένωσης. Και είδαμε δυστυχώς στις 25 Μαΐου πως αυτή η αναγνώριση δεν είναι κάτι κεκτημένο. Εάν η Ευρώπη δεν μπορεί να ολοκληρώσει ε, αισίως προγράμματα που έχουν ε, αντίκτυπο επιτόπου, στο τοπικό επίπεδο, δεν θα γίνει αντιληπτό λοιπόν αυτό. Ήδη παλιότερα μιλούσαμε για έναν προπολογισμό ε, της τάξης του 1,24% του ΑΕΠ. Τώρα πόρο απέχουμε από αυτό. Είμαστε στο 1% στις πιστώσεις ε, υποχρεώσεων και στο 0,94% για το πληρωμές. Ε, τι θα πει αυτό, οι υποχρεώσεις αναλαμβάνονται για να δουλέψουμε σε διάρκεια. Ε, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν πιστώσει πληρωμών που να είναι τουλάχιστον αντίστοιχε. Εφόσον να υπάρχουν τέτοιο επιπέδου διαφορέ, σημαίνει ότι στην ουσία κάνουμε ε, ό,τι να είναι. Γιατί Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα που είναι ουσιαστικό και είναι αλήθεια ότι για τα ε, εδάφη και είμαι πρόεδρος μιας ε, ε, γαλλικής περιφέρειας για τα τοπικό επίπεδο δηλαδή, τα διευθυντικά ταμεία και ο αντίκτυπός τους είναι πολύ σημαντικά. Παίζουν ρόλο μοχλού για διάφορες δημόσιες πολιτικές, δηλαδή χωροταξία, υποδομές, παιδεία, κατάρτιση, ένα σωρό θέματα που άμεσα ενδιαφέρουν το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών και πιστεύω πως σήμερα δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε να μας ε, κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να αντισταθούμε σε σχέση με τα όσα προτείνει το Συμβούλιο και να εξηγήσουμε πως είναι προς το συμφέρον του ίδιου του Συμβουλίου και των κρατών να είναι πιο ορατή, πολύ πιο ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες και το έχουμε πει και ξαναπεί στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, ότι το θέμα των ιδίων πόρων θα πρέπει να μας απασχολήσει κατά προτεραιότητα στην Επιτροπή μας, γιατί αν συνεχίσουμε να κάνουμε τα πηγενέλα ανάμεσα στο τι δίνουν τα κρατημέλη και στο τι παίρνουν πίσω κτλ, δεν θα λειτουργήσουμε ικανοποιητικά. Πρέπει λοιπόν πολύ γρήγορα να εγγύψουμε στο θέμα των ιδίων πόρων, ιδιαίτερα στην φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κόρνελ για την τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο εισηγητρίες. Νομίζω ότι σαφές από όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν ποια είναι η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα και εγώ να μεταφέρω τη δική μου θέση. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο μας θα πρέπει να αγωνιστεί για να υπάρξει πραγματικά αξιόπιστος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφαρμόζεται σωστά. Συγκεκριμένη όμως αυτή η περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο των πιστώσεων υποχρεώσεων και το ε, ποσό των πιστώσεων πληρωμών θα πρέπει να είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα χάσμα το οποίο δημιουργείται και το οποίο διευρύνεται από το ένα χρόνο στον άλλο και η δική μου εντύπωση είναι ότι κανείς δεν μπορεί πια να προβλέπει πότε θα μπορέσουν να γίνουν οι πληρωμές των υποχρεώσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν και κανείς δεν ελέγχει ποιος αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεν θα πληρωθούν. Αυτό δεν οδηγεί σε καμία διαφάνεια έναντι των πολιτών και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τη δυνατότητα δράσης. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε τον έλεγχο των υποχρεώσεων που συνάπτονται εξίσωση βέβαια των πιστώσεων πληρωμών με τις πιστώσεις υποχρεώσεων, αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξηθεί αυτομάτω. Γιατί οι πολίτε μα δεν θα το καταλάβουν αυτά. Τα χρήματα αυτά δεν είναι δικά μα χρήματα, είναι χρήματα των φορολογουμένων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή διαχείριση σε αιτήσιο επίπεδο και να μην δημιουργούνται αποθεματικά τα οποία είναι πλασματικά αποθεματικά, γιατί ξέρουμε ότι πολλέ φορέ τα αποθεματικά αυτά είναι μονάχα για να δαπανηθούν σε συγκεκριμένου τομεί. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί και καλύτερο σχεδιασμό στα θέματα αυτά. Συμπεραίνω ότι χρειαζόμαστε ένα πλήρε πλαίσιο και ένα σαφέ πλαίσιο για τι πληρωμέ μα και μόνο με αυτή τη βάση μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Θα ήθελε να παρέμβει η Κομισιόν. με τον που έχει εδώ παρόντα το Γενικό Διευθυντή του Προϋπολογισμού. Ε, θα ήθελα να κάνει κάποια σχόλια. Έχετε το λόγο κυρία Γενική Διευθυντή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι προς το παρόν η Κομισιόν χαιρετίζει τα σχόλια των βουλευτών. Έχουμε ακούσει με μεγάλη προσοχή τη θέση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσβλέπουμε στη συνεργασία με την Επιτροπή σας. Όπως ε, τονίσατε είναι σημαντική η διαφάνεια και η σαφήνεια για να έχουμε μια συμφωνία ή δυνατόν το φθινόπωρο. Πολύ ωραία. Με κάπως περισσότερες πληρωμές ενδεχομένως λέει ο πρόεδρος και κάπως λιγότερες πιστώσεις υποχρεώσεων. Δεν ξέρω αλλιώ μπορούμε να έχουμε κάποια λύση. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω στις δύο εισηγήτριές μας, τη Γενική Εισηγήτρια και την εισηγήτρια για το τμήμα 3 να μας δώσουν τα συμπεράσματα που αντλούν από αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Βλέπω ότι τα μέλη της Επιτροπής μας που έλαβαν το λόγο βρισκόμαστε όλοι στην ίδια οδική γραμμή. Πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα αυτό των πιλωτών, των πληρωμών. Αλλά Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα. Δεν είναι μονάχα μια διαλκυστίνδα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Δεν είναι μια μάχη για να έχουμε μια διαμάχη. Υπάρχει ένα πραγματικά φιλοσοφικό πρόβλημα. Ο στόχος του προπολογισμού θα πρέπει να είναι να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στους τομείς που εμείς θεωρούμε ότι είναι τομείς προτεραιότητες. Και πάντα υπάρχει η έννοια της προσθέμενης αξίας που πρέπει να ε, πριτανεύει στην περίπτωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Βέβαια, αυτό εφόσον καταβληθούν οι πληρωμές, γιατί χωρίς πληρωμές δεν υπάρχει ούτε προσθέμενη αξία, αλλά ούτε αξιοπιστία, ούτε τόνωση της οικονομίας. Εδώ δώσαν οι συνάδελφοι τα παραδείγματα μιας περιφέρειας ή μιας ε, δημοτικής αρχής που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά δεν παίρνουν ανάκτηση των κονδυλίων που καταβάλουν για αυτά τα προγράμματα. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και υπάρχουν και άλλα θέματα όπως το θέμα των πληρωμών για, το έρασμο, για τον έρασμο που είναι ένα πολύ συμβολικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ο κόσμος να συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να υπάρχουν ανθρωπιστικά προγράμματα όπου συμμετέχουν ΜΚΟ παραγματικά χάρη ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν εύκολα και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και μετά καθυστερούμε να τους δώσουμε τις πληρωμές τους. Δεν είναι λοιπόν θέμα αριθμών, δεν είναι θέμα διαθεσμικής διαμάχης. Το θέμα είναι ότι εμείς θέτουμε αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο τον, την προσθέμενη αξία που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Γι' αυτό ζητώ κατηγορηματικά να υπάρξει υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων και να κρατήσουμε μια στεναρή θέση στις διαπραγματεύσεις έναντι του Συμβουλίου. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια ομοφωνία μεταξύ μας και μια γενική συνέντευξη για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε σωστά με το Συμβούλιο. Θα τα καταφέρουμε στο τέλος που θα πάει. Ε, παρακαλώ κύριε Χολμάγερ. Μόνο κι εγώ ένα σχόλιο θέλω να κάνω για τον προπολογισμό της Κομισιόν. Είναι πράγματι δύσκολο. Να βλέπουμε συνέχεια το Συμβούλιο το οποίο ουσιαστικά παραβαίνει τις δικές του αποφάσεις και δεν δέχεται να πληρώσει τις ε, υποχρεώσεις που έχει συνάψει. Πρέπει λοιπόν εμείς να βρούμε ε, και εμείς ποιες πρέπει να είναι οι δικές μας προτεραιότητες μαζί με την Κομισιόν να δούμε ποιοι είναι ακριβώς οι τομείς οι οποίοι θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητες. Δεν είναι εύκολο αυτό να πούμε ότι σε κάποιους τομείς θα πρέπει να παραμελήσουμε τις πληρωμές και αλλού να τις ενισχύσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έχουμε μια τέτοια ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Επανέρχομαι τώρα στα θέματα του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ουσιαστικό γιατί καταφέραμε να έχουμε μια κοινή πορεία με τον, ε, το, προηγου, με το Προεδρείο κτλ. Και φυσικά υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα της Επιτρόπης Περιφερειών που προανέφερα και το πρόβλημα του δικαστηρίου όπου υπάρχει πραγματικά μια δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπιστεί και εξάλλου έχουμε και μια δύσκολη κατάσταση σε σχέση με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και τη υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά για το δικαστήριο κυρίως είναι απόλυτα αδύνατο να αποδεχθούμε ε, την κατάσταση αυτή που δημιουργείται από το Συμβούλιο και επειδή είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό του χρηματοδότηση του δικαστηρίου σε σχέση με το γενικό προπολογισμό, είναι τελείω απαράδεκτο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Γενική Συγγήτρια και την Συγγήτρια του Τμήματο 3. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλε σα τι διευκρινήσει. Από την σημερινή ανταλλαγή απόψεων πρέπει να εμπνευστείτε, να νιώσετε ότι έχετε τη στήριξη όλων όσοι πήραν το λόγο. Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε σε μια τέτοια αμφίσιμη κατάσταση. Δεν μπορεί, είναι προσβλητικό να μένουν απλήρωτοι λογαριασμοί, προσβλητικό για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει συγχρόνως να, να θυμίσουμε σε όλους τους ε, συναδέρφους ότι οι υποχρεώσεις είναι ένα πράγμα, αλλά να δεν ακολουθούν και οι πληρωμές, ανάλογα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είμαστε λοιπόν στην αρχή αυτής της θητείας και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα αποφασισμένοι να διευθετηθεί το θέμα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον προπολογισμό του 2015, σχέδιο προπολογισμού για την κινητοποίηση, ευελιξία, αλληλεγγύη κλπ. Δεν έχουμε εισηγητή, θα επανέλθουμε λοιπόν αρχές Σεπτεμβρίου. Και έτσι Τώρα περνάμε στο 2014. Διορθωτικός προϋπολογισμός, αριθμός 2, 3 και 4. Ο εισηγητής μας λοιπόν, ο Ζεράρ Ντεπρέ παρακαλώ να μας παρουσιάσει τα τρία αυτά σχέδια διορθωτικού προϋπολογισμού. Και θέλω να πιστήσω εδώ την προσοχή σας και στο εξή. Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθμός 3 έχει να κάνει με το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης που είναι η κινητοποίηση του αποθεματικού για τα πρόβλεπτα. Εδώ δεν έχουμε ακόμα εισηγητή. Αυτά τα τρία σχέδια προπολογισμού έχουν βέβαια διαφορετικές επιπτώσεις στους αναγκαίους πρόσθετους πόρους. Ενώ το σχέδιο προπολογισμού 3 ανεβάζει στα 4 δις 700 εκατομμύρια, Παρόλα αυτά χρειαζόμαστε επιπλέον ε, πόρους από το απόθεμα που εμφανίζεται στο σχέδιο προπολογισμού 2 και ο κύριος Ντεπρέ έχει το λόγο για να μας τα εξηγήσει αυτά λεπτομερέστερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, το είπατε και εσείς, θα σας παρουσιάσω συγκεντρωμένα το 2, 3 και 4. Και δεν θα σας τα παρουσιάσω απλώς συγκεντρωμένα όλα αυτά, αλλά θα κάνω και την πρόταση να τα εξετάσουμε έτσι και τα τρία μαζί όταν θα έχουμε διαπραγματεύσεις επ' αυτού με το Συμβούλιο. Η πρόταση αυτή για να τα εξετάσουμε μαζί αυτά τα τρία σχέδια προπολογισμού ήταν μια πρόταση που έκανε ο προηγούμενος Γενικός Εισηγητής για το 2014 που ήταν η κυρία Γένσεν. Εμείς το στηρίξαμε στον τριμερή διάλογο που είχαμε, αν δεν απατώμε 10 Ιουλίου. Και στην σημερινή συνεδρία σήμερα το πρωί οι συντονιστές των διάφορων πολιτικών ομάδων συμφώνησαν με αυτή την αντιμετώπιση. Συνεπώς πρόκειται για τρία σχέδια διορθωτικών προπολογισμών που παρουσιάζονται και θα στηριχτούν από εμά στο Συμβούλιο. Όσον αφορά το καθένα από τα σχέδια αυτό, να σας κάνω πρώτα μια γενική παρουσίαση για το σχέδιο αριθμός 2. Εδώ πρόκειται για το απόθεμα που έχουμε από το 2013, το οικονομικό του 2013. Και όσον αφορά τα έσοδα και όσον αφορά τις δαπάνες πρόκειται για ένα δισεκατομμύριο, 500 εκατομμύρια ευρώ και κάτι ψηλά. Δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα, έχει ήδη εγκριθεί ουσιαστικά από το Συμβούλιο. Εγκρίνοντά το βέβαια, το Συμβούλιο και δεν ξέρω αν αυτό το έχει καταλάβει, δημιουργεί τι προποθέσει ώστε διάφορε χώρε μέλη να μπορούν να πάρουν μια επιταγή επιστροφή από την μη χρήση μέρους των προπολογισμών που είχαν καταγραφεί, των κονδυλίων που είχαν καταγραφεί. Έχω να κάνω εδώ την εξή πρόταση. Στην περίπτωση που θέλουμε να εξετάσουμε μαζί με το Συμβούλιο το 2, το 3 και το 4, θα πρέπει, είναι αναγκαίο θα έλεγα, να προτείνουμε μία αλλαγή στο 2 για να είμαστε σίγουροι ότι συγκλίνουν τα χρονοδιαγράμματα ανάμεσα στο σχέδιο 2 που έχει ήδη εγκρίνει το Συμβούλιο και το 3 και τα 4 που ακόμα δεν έχουν εγκριθεί. Συνεπώς πρέπει να αποφανθούμε και επί μια τέτοια τροπολογίας που είναι σημαντική δεδομένου ότι το πολιτικό βάρος είναι μεγάλο. Το δεύτερο τώρα σχέδιο διευθυντικού προπολογισμού αριθμός 3. Αυτό είναι κάπως πιο επίμαχο, πιο λεπτό το Συμβούλιο εδώ ζητά επιπλέον πιστώσεις για 4 δισεκατομμύρια 738 εκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών. Είμαστε στις πληρωμές λοιπόν τώρα. Επιπλέον πιστώσεις 4 δισεκατομμύρια 738 εκατομμύρια. Το ποσό μειώνεται με τις με μείον τις επιπλέον δαπάνες προστίθεται στο 2014. Πρόκειται δηλαδή για το 3, 3 εκατομμύρια 3 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια. Τελικά καταλήγουμε αφαιρώντας τα πλεονάσματα κτλ. Αυτές τις επιπλέον λοιπόν πιστώσεις πρέπει να τις πληρώσουμε. Είναι μια διπλή πρόταση αυτή. Γιατί πρώτον λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μη χρησιμοποιημένο περιθώριο για την οροφή των πληρωμών 700 εκατομμύρια περίπου. Και δεύτερον πρόκειται για την ε, μετακίνηση του περιθωρίου για τα πρόβλεπτα. 4 εκατομμύρια. Το 4 δις εδώ. Κανονικά έχουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 0,030% κανονικά Και εδώ είναι που κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν σημαντικές δυσκολίες με το Συμβούλιο στην περίπτωση που κάποιες χώρες μέλη έχουν πει πως η κινητοποίηση αυτού του μέσου δεν δικαιολογείται. Έρχομαι τώρα και στο σχέδιο 4 και τις προτινόμενες αλλαγές επιπλέον έσοδα. Όπως Είπατε, εδώ πέρα πρόκειται για καθυστερημένες πληρωμές, 2 δισεκατομμύρια 59, που οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι οι επιθωρήσεις δεν θα γίνουν τότε που είχαν προβλεφθεί, οπότε οι επιπλέον δαπάνες δεν προλαβαίνανε να γίνουν. 2 δισεκατομμύρια, 59 εκατομμύρια λοιπόν είναι λιγότερο το ποσό που χρειάζεται. Συνολικά λοιπόν, το απόθεμα από την χρήση 2013 1 δισεκατομμύριο ευρώ 4 δισεκατομμύρια 738 από, τις επιπλέον, τα επιπλέον έσοδα στο 3 και στο 4 συνεπώς μας μένει ένα πλεόνασμα να καλύψουμε 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν εδώ βάλουμε μαζί τις τρεις αυτές προτάσεις για διορθωτικό προϋπολογισμό, αυτό σημαίνει ότι δεν δίνουμε πίσω στο Συμβούλιο στις χώρες μέλη δηλαδή το ποσό που έχουμε πλεόνασμα από το 2013 βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού 2, αν λάβουμε υπόψη μας το πλεόνασμα αλλά και, τις επιπλέον, ε, και τα επιπλέον έσοδα που έχουμε από το 3 και το 4, μένουν 105 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει 105 δισεκατομμύρια ευρώ. 105 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι λοιπόν το περιθώριο που έχουμε για τα πρόβλεπτα, που είναι πέρα από τις επιτρεπόμενες πληρωμές ήδη και αυτή ακριβώς είναι και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπάρχει στο επόμενο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Προτείνω λοιπόν, Πρόεδρε, να συμφωνήσουμε με τις τρεις αυτές προτάσεις που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις δούμε συνολικά, να τις υποστηρίξουμε στο Συμβούλιο συνολικά, να εισάγουμε και μία τροπολογία για τον διορθωτικό προπολογισμό αριθμός 2 για να υπάρχει συνοχή στο χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και να μην κάνουμε πίσω. Αν αυτές οι πιστώσεις πληρωμών επιπλέον για τη χρήση 2014 είναι αναγκαίες για τον προπολογισμό 2014-2015. Αν δεν γίνει αυτό, τότε ο προπολογισμό του 2015 θα επιβαρυνθεί επιπλέον για τι πληρωμέ. Αυτά είχα να πω προ το παρόν, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ για αυτή τη ε, διαφωτιστική εισήγηση. Θα μειωθούν ε, κάποια δι ε, τα, τα χρωστούμενα. Η κυρία Γενική Συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που είπε μόλις τώρα ο κύριος Ντεπρέ, δηλαδή να είναι συνολικό το πακέτο αυτό των τριών διορθωτικών προπολογισμών, γιατί έτσι καλλιώς πρόκειται για πληρωμές και στις τρεις περιπτώσεις, έτσι καλώς είναι αυτά τα τρία είναι απόλυτα λογικό λοιπόν κατά τη γνώμη μας να εξεταστούν από κοινού οι διορθωτικοί αυτοί προπολογισμοί. Επιπλέον, επειδή βάζοντας και τους τρεις μαζί, η πρόταση τελικά που κάνουμε στο Συμβούλιο γίνεται έτσι πιο εύπευτη, είναι πιο εύκολο το Συμβούλιο να την αποδεχτεί από ότι αν παρουσιάζουμε για παράδειγμα χωριστά το διορθωτικό προπολογισμό 3, ξέροντας τις ε, θέσεις που υποστηρίζουν οι χώρε μέλη θα ήταν δύσκολο να το δεχτούμε. Οπότε αυτό είναι καλό. Εμείς χρειαζόμαστε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή γιατί ξέρουμε ποια είναι τα πρόστιμα. Οπότε το Συμβούλιο αυτό που προτείνει είναι τι, τίποτα. Να μην υπάρχουν ε, παραπάνω χρήματα και αν υπάρχουν να είναι μόνο για μέρος των λογαριασμών. Θέλω επίσης να πω κι εγώ όπως έλεγε και ο κύριος ο ηγητής μας, ότι δεν είναι δυνατόν τις διαπραγματεύσεις για το προπολογισμό 2015 να τις ξεκινήσουμε αν δεν έχει λυθεί ή εν πάση περιπτώσει αν δεν έχει μπει ένα φιλοπορίας κατά κάποιο τρόπο για ό,τι μας μένει μέχρι τώρα. Γιατί το επίπεδο των πληρωμών που χρειαζόμαστε για το 2015 θα, εξαρτηθεί από τον προπολογισμό 2014 και από το τι εκρεμεί από τις προηγούμενες χρονιές. Όσο λοιπόν δεν υπάρχει συμφωνία για τους διορθωτικούς αυτούς προπολογισμού και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση των πληρωμών στις 31 Δεκεμβρίου, για να το πω έτσι, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ποιες θα είναι και οι ανάγκες μας για το 2015. Διότι οι προϋπολογισμοί δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, δηλαδή να είναι όλοι μεμονωμένοι και ο καθένας να έχει τις προβλέψεις και τα δικά του τα ποσά, αλλά επειδή μας μένουν απλήρωτοι λογαριασμοί από τις προηγούμενες χρονιές, πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Προέδρο, ευχαριστούμε πολύ κυρία Γενική Συγκητρία. Ωραία, βλέπω ότι συμφωνείτε με τον κύριο Ντεπρέ όσον αφορά το πακέτο και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα τη διόρθωση 2014 και τον προπολισμό του 2015. Σχόλιο παρακαλώ. Δεν βλέπω σχόλια. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. Παρακαλώ. Α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω τέσσερα σχόλια σε σχέση με τον με τη συζήτηση του σχεδίου διορθωτικού προπολογισμού. Πρώτα απ' όλα, να σα εξηγήσω τον ε, διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 3 που ανέφερε ο κ. Στεπρέ, ο οποίο είναι και πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά τα ποσά και σε ό,τι αφορά το γεγονό ότι έχει να κάνει με δάπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ήθελα να σα εξηγήσω ότι η Κομισιόν πρότεινε αυτό τον ε, διορθωτικό προπολογισμό ω πράξη ευθύνη. Είδαμε ότι είχε προχωρήσει πολύ η εφαρμογή των προγραμμάτων ήδη από την Άνοιξη. Τώρα Συνεχίζει η εφαρμογή των προγραμμάτων. Έχουμε φτάσει στα 70% απορρόφηση των κονδυλίων και τα πράγματα έχουν προχωρήσει προς την κατεύθυνση ενός προβλήματος ως το τέλος του χρόνου. Έχουμε χρησιμοποιήσει δύο εργαλεία σε αυτό το διορθωτικό προϋπολογισμό. Καταρχήν χρησιμοποιούμε το περιθώριο 700 εκατομμυρίων που υπάρχει για τις πληρωμές και τα 4 δισεκατομμύρια για το αποθεματικό ε, εκτάκτων αναγκών. Επίσης, ε, αυτό που ανέφερε ο κύριος Ντεπρέ, όταν η Κομισιόν εξέφρασε την απόψή της ότι συμφωνεί για το πολιετές πλαίσιο δημοσιονομικών δαπανών, είπαμε ότι θα μπορέσει να είναι λειτουργικό αυτό το πλαίσιο και να εφαρμοστεί αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα περιθώρια ευκαμψίας που περιείχονται στο σύστημα. <clears throat> Υπήρξε λοιπόν και μια συμφωνία με τα δύο σκέλη της αρχής του προπολογισμού ότι ήταν απαραίτητη αυτή η ευκαμψία για την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Η ευκαμψία υπάρχει σε διάφορα εργαλεία. Ένα είναι το πλαίσιο αυτό ε, ερεσιμότητος, το οποίο μας επιτρέπει να δώσουμε κονδύλια πιο νωρίς από ό,τι προβλέπετε. Επίσης υπάρχουν άλλα εργαλεία τα οποία είναι ad hoc και τα οποία επιτρέπουν να ξεπεράσουμε τις οροφές και τις πληρωμές. Ένα άλλο στοιχείο ευκαμψίας είναι το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού που πρέπει να το πράξει η Κομισιόν, να το προτείνει η Κομισιόν για να λάβουμε υπόψη τις ε, απρόβλεπτες ταπάνες οι οποίες μπορούν να προκύψουν, πολλές φορές είναι αρνητικού χαρακτήρα πρόσθετα στοιχεία δαπανών, μερικές φορές είναι και θετικά νέα, δηλαδή πρόσθετα απρόβλεπτα έσοδα. Μπορεί πράγματι να αλλάξει η κατάσταση και μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το <clears throat> πώς πηγαίνει η απορρόφηση των κονδυλίων του προπολογισμού, παρά το γεγονό ότι Σεπτέμβριο θα ξέρουμε ακόμα καλύτερα για τι πιστώσει πληρωμών, αλλά μπορεί να υπάρξουν και πρόσθετε δαπάνε οι οποίε θα προελθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύη και εδώ πρέπει να σα προειδοποιήσω και ενδεχομένω θα υπάρχουν και θετικά νέα γιατί μπορεί παραδείγματο χάρη να μην υπάρξουν ε, ενστάσεις και προσφυγές από εταιρείες στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα λάβουμε υπόψη για να έχουμε ένα ρεαλιστικό τρόπο εφαρμογής του προϋπολογισμού. Τρίτο στοιχείο, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Τεπρέ, το φθινόπωρο θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση του αν θα χρησιμοποιήσουμε το πρόσθετο, τα πρόσθετα έσοδα που έχουμε για να πληρώσουμε τα οφειλόμενα ή όχι. Κατά τη δική μου άποψη είναι απόλυτα λογικό, επειδή έχουμε πολύ υψηλά κονδύλια τα οποία έχουν μείνει απλήρωτα, να χρησιμοποιήσουμε τα πρόσθετα έσοδα για να πληρώσουμε αυτά τα οφειλόμενα, ώστε να μην συνεχίσουν τα, υπο, τα μη εκταμιευθέντα ποσά να αυξάνονται. Τέλος, τελική μου παρατήρηση. Θέλω να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε ο κ. Λεβαντόφσκι, ο κ. Δεπρέ και άλλοι. Μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Λεβαντόφσκι, ο οποίος ήταν επίτροπος για τα θέματα του προπολογισμού μέχρι πρόσφατα, <clears throat> για τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 3 και για την διαρρύθμιση των πληρωμών το 2014 να γίνει πιο λογικά πρέπει να γίνει πιο αξιόπιστος ο προϋπολογισμός του 2015. Είναι ο δεύτερος μέσα στο νέο πολιετές πλαίσιο και έχει μερικά θετικά στοιχεία σε σχέση με το εφετινό προϋπολογισμό. Όχι μόνο πληρώνουμε τα οφειλόμενα του παρελθόντος, αλλά ξεκινάμε νέα προγράμματα και ξεκινάμε την εφαρμογή του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και αυξάνεται, διπλασιάζεται ουσιαστικά το ποσοστό των ποσών που πληρώνονται για τα νέα αυτά προγράμματα. Εάν θέλουμε ο προπολογισμό του 2015 να συμβάλλει πράγματι στο να βγει η Ευρώπη από την κρίση, θα πρέπει να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τις πληρωμές το 2014, ώστε να μην αντικαταστήσουμε μια, αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου οι πληρωμές το 2015 θα είναι ουσιαστικά πληρωμή οφειλωμένων από το παρελθόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γενική Διευθύντρια για τα αισιόδοξα σας σχόλια μπορεί να έρθει και ο Άι Βασίλης από το καλοκαίρι και να μας βοηθήσει ήδη. Και θα ήταν πολύ καλό να φύγουμε διακοπές με αυτή τη θετική προοπτική. Ούτως ή άλλως, είπατε ότι πρέπει να, είναι σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των πληρωμών, εφόσον έχουν αναλυφθεί υποχρεώσεις, πρέπει να καταβληθούν και οι πληρωμές. Αυτά λοιπόν <clears throat> για το 2014. Και τώρα έχουμε την κινητοποίηση του περιθωρίου ερεσιμότητος, ο κύριος Δεπρέ. Φοβάμαι κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό αρκετά γρήγορα. του περιθωρίου για τις απρόβλεπτες ανάγκες. Είναι απαραίτητο να κινηθούμε γρήγορα για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τον προπολογισμό το διορθωτικό υπαριθμών 3. Θα ήταν λοιπόν ε, χρήσιμο να το κάνουμε το ταχύτερο. Αν κανείς άλλος δεν ενδιαφέρεται θα μπορούσα εγώ να είμαι εισηγητής για αυτό το θέμα γιατί πραγματικά με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα του διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 3 και δεν έχουμε κανένα συμφέρον να καθυστερούμε την έγκριση αυτού του νέου προπολογισμού. Ο διορισμός τώρα εισηγητή για τις απρόβλεπτες δαπάνες είχαμε αποφασίσει να οριστεί ο εισηγητής για, για το Ταμείο Προβλέπτων Δαπανών το Σεπτέμβριο. Δεν έχω πρόβλημα, λέει ο κύριος Σέντεπρε. Εγώ θα ήθελα να γίνει το ταχύτερο δυνατό η έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού και αυτό προϋποθέτει το διορισμό εισηγητή ώστε να μπορέσει να εκτελεστεί αυτός ο προϋπολογισμός. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Και αυτό που λέτε δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε το αργότερο στις 3 Σεπτεμβρίου να ορίσουμε εισηγητή και να επιτρέψουμε στον εισηγητή αυτό να εκφράσει την απόψή του το ταχύτερο δυνατό. Όσοι είναι υποψήφοι για αυτή τη θέση πρέπει να το γνωρίζουμε Μπορούμε τώρα να περάσουμε την ε, κινητοποίηση του Ταμείου προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι τα σημεία 10 με 14. Και εδώ υπάρχει το ίδιο χρονοδιάγραμμα. Και επομένως μπορώ να δώσω το λόγο διαδοχικά στους εισηγητές και μετά μπορεί να υπάρξει μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Ίσως αυτό είναι καλύτερο από το να τα συζητήσουμε και τα πέντε θέματα από κοινού. Η EGF 2014-01 Nutriart, ο κύριος Κίρτσος έχει το λόγο.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 Οι ελληνικές αρχές ε, κατέστησαν υποχρεωτικό το Φεβρουάριο 2014 να, δίνεται, να δοθεί ε, μια οικονομική βοήθεια για, από το Ταμείο Προσαρμογής στην ε, Παγκοσμιοποίηση μετά από απολύσεις από την εταιρεία Nutriart και μικρότερες εταιρείες. Η Nutriart είναι η πιο μεγάλη και σημαντική το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, το EGF, θεσπίστηκε για να δώσει στήριξη στου εργαζόμενου που απολύονται αλλά και στου ανεξάρτητους επαγγελματίε, των οποίων η δραστηριότητα έχει πάψει λόγω μεγάλων διαθετικών αλλαγών στα παγκόσμια σχήματα εμπορίου, λόγω παγκοσμιοποίηση αλλά και λόγω των συνεπειών τη παγκοσμίου οικονομική κρίση. Η Νούτρι Άρτε ήταν μια ε, φημισμένη εταιρεία στην Ελλάδα έπαυσε τις λειτουργίες της, έφτιαχνε ειδικά είδη ψωμιού, δημητριακά, μπισκότα και ήταν παρούσα στην χώρια αλλά και στη διεθνή αγορά. Θα πρέπει να πούμε πως η Κομισιόν αντέδρασε ταχύτατα και αποτελεσματικά εφόσον ε, μέσα σε περίοδο τεσσάρων μηνών δημοσίευσε την αξιολόγησή της για την υπόθεση Νουτριάρτ. Η Κομισιόν ολοκλήρωσε σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ότι οι προϋποθέσεις για την παροχή οικονομικής βοήθειας από την, ε, το Ταμείο αυτό ε, πληρούνταν. Και γι' αυτό και έκανε πρόταση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η αίτηση αφορά 508 εργαζόμενους της Nutriart καθώς και άλλες εταιρείες που είχαν σχέση με την Nutriart είναι περίπου 25 ε, ανεξάρτητους επαγγελματίες που επίσης έχασαν την ε, δραστηριότητά τους. Οι ελληνικές αρχές ε, προσφέρουν προσωπικές ε, ε, υπηρεσίες σε 505 νεαρούς με απασχόληση, κατάρτιση, ε, η μαθητεία, νέος που είναι κάτω από την ηλικία των 30, γιατί οι απολύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 συνέβησαν στην ε, περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, Αττική, ε, ευρύτερη περιοχή Αθηνών δηλαδή, και πρόκειται για περιοχές που είναι επιλέξιμες σύμφωνα υπό την μάλλον πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Πρόκειται λοιπόν για 113 ε, ανθρώπους ε, που θα υποφεληθούν. Η Θεσσαλονίκη και Αθήνα είναι οι μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας. Το μέσος όρος ανεργίας σε εθνικό επίπεδο είναι 26 με 27% του εργατικού δυναμικού ίσως να είναι, είναι σίγουρα ευρωπαϊκό, ίσως και παγκόσμιο ρεκόρ το ποσοστό αυτό. Οπότε χρειαζόμαστε αυτές τις προσπάθειες από πλευράς της των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και επίσης οι δικαιούχοι θα βοηθηθούν μέσω επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης, μαθητείας ε, συμβουλευτικών διαδικασιών, καθώς και ειδικέ ε, επιδοτήσεις για τη δημιουργία ιδιωτικής επιχείρησης, αλλά και για την κινητικότητα. Είναι μια προσπάθεια να αυξηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων και να δοθεί μια ευκαιρία στον κόσμο αυτό να επανέλθει, να επανενταχθεί εργατικό δυναμικό σε πολύ δύσκολες κοινωνικές συνθήκες. Το σύνολο των χρημάτων που ζητούνται από το ETF, EGF είναι 6.096.000 ευρώ, που είναι το 60% του συνολικού κόστους. Οι ελληνικές αρχές υπέδειξαν ότι η οικονομική βοήθεια του Ταμείου δεν θα αντικαθαστήσει δράσεις που είναι υποχρεωτικές για τις εταιρείες αυτές με βάση την εθνική νομοθεσία ή απορρέουν από συλλογικές συμβάσεις. Η εθνική προχρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση είναι το, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη. Οι ελληνικέ αρχέ επίση υπέδειξαν πω τα μέτρα που περιγράφονται εδώ και που θα λάβουν οικονομική βοήθεια από το EGF δεν θα λάβουν οικονομική βοήθεια από άλλα ταμεία της κοινότητας. Τώρα, για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Κομισιόν υπέβαλε στις δημοσιονομικές αρχές ένα αίτημα μεταφοράς για ένα συνολικό ποσό 6.096.000 ευρώ από το αποθεματικό του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, μεταφορά δηλαδή από το Ταμείο στην αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού. Πρόταση μεταφοράς για την κινητοποίηση του Ταμείου που έχει διαβιβαστεί ε, μέσα στο 2014. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την αξιολόγηση και την θέση της Κομισιόν, γιατί ε, η χώρα μου βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Η ελληνική οικονομία έχει πάψει να μειούται. Έχουμε χάσει το 25% του ΑΕΠ μας από το 2008 μέχρι σήμερα και υπάρχουν κάποια σημάδια ανάκαμψης. Αλλά υπάρχει μεγάλο χρονικό μεγάλη χρονική απόσταση ανάμεσα στα ίχνη, αυτή, ίχνη αυτά της ανάκαμψης και την απασχόληση που έχει φτάσει σε υψηρή κόρο. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν σχόλια. Ε, ε μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι νέο μέλος αυτής της Επιτροπής και είμαι επίσης και μέλος στην Επιτροπή Απασχόλησης όπου υπάρχει μια ομάδα εργασίας για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και είχαμε μια συζήτηση με την Κομισιόν για τα θέματα αυτά και εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση προς τον εισηγητή που μπορεί να ενδιαφέρει και τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Είναι η πρώτη περίπτωση όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό για την εκπαίδευση και την ε, κατάρτιση των νέων και είχαμε χθε μια συζήτηση στην ομάδα εργασίας για το αν στην περίπτωση αυτή ε, έχει υπάρξει μια σωστή εφαρμογή αυτού του συστήματος και γι' αυτό θα είναι χρήσιμο να αποκομίσουμε τις εμπειρίες από αυτή την περίπτωση για το πώς στη συνέχεια θα μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Δεν θέλουμε λοιπόν αυτό να αφαιθεί μονάχα στα χέρια των κρατών μελών. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει πολύ θετικέ συνέπειε για του νέου. Είναι κάτι που πρέπει να υποστηρίξουμε. Πρέπει να υποστηριχθεί λοιπόν η απασχόληση των νέων, αλλά θα πρέπει να είναι πιο σφιχτή η διαδικασία για την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Και θα ήθελα λοιπόν να τα μεταφέρω όλα αυτά στην Επιτροπή μας, γιατί είναι μια πρώτη περίπτωση που γίνεται εφαρμογή αυτού του συστήματος. Merci, σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις σα, κυρία Γκρέσλε. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο έχει κάνει μια έκθεση για τα θέματα αυτά, μια ειδική έκθεση για το Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Ο Βίλι Ήταλε, ο παλιός συνάδελφός μας ήταν αυτός ο οποίος είχε καταρτήσει αυτή την έκθεση και ίσως θα έπρεπε να τον καλέσουμε να την παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής μας. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και μπορούμε να αποκομίσουμε πολλά διδάγματα από αυτήν. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, κυρία Γκρέσλα. Στο τέλος της συνεδρίας θα το ανέφερα το θέμα αυτό. Ήταν, θα είναι χρήσιμο να σκεφτούμε λοιπόν και για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε αλλά ενδεχομένω μαζί σας με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ε, <clears throat> εκθέσεις αυτές του ελεκτικού συνεδρίου που μας δίνουν σημαντικές ε, πληροφορίες για το πράκτο Ο κύριο Κολμέλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει γενική συμφωνία ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι να μπορέσουν να αποκομίσουν μια θέση εργασία. Εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί βέβαια, να μην έχουμε μονάχα ένα τίτλο ο οποίος θα παρουσιάζεται. Πρέπει να έχουμε και ουσία πίσω από τον τίτλο. Στο συγκεκριμένο αυτό το τομέα της ε, απασχόλησης των νέων θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι πράγματι μόνιμου χαρακτήρα και όχι μονάχα ότι δίδεται μια αρχική ε, βραχυπρόθεσμη λύση η οποία στην πράξη δεν πρόκειται να αλλάξει σε τίποτα και δεν πρόκειται να βελτιώσει τις δομές. Ιδίω για αυτά τα προγράμματα αυτά, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε να υπάρχει μια αξιολόγηση για να ξέρουμε τι προήλθε από αυτά τα προγράμματα και να μπορέσουμε να διδαχτούμε και αυτά τα προγράμματα με τον, για, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε μελλοντικά να τα βελτιώσουμε. Για αυτήν την περίπτωση φυσικά δεν μπορώ να πω ακόμα τίποτα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να λάβει τον λόγο. Σας υπενθυμίζω ότι θα επανέλθουμε στην συνεδρίασή μας στις 11 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να εγκριθεί στην Ολομέλεια στις 16 Σεπτεμβρίου. Και αυτό αφορά και τις άλλες αιτήσει κινητοποίησης του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Και έχουμε τώρα την πρόταση για τεχνική βοήθεια με, πρωτοβουλία της Κομισιόν ΤΑΦ Α2014. Και εγώ συμφωνώ με τα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί να χρηματοδοτηθούν ως τεχνική βοήθεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα διευκολύνει την ε, ε, εκταμείευση των τομέων των ε, κονδυλίων αυτών και υποστηρίζω και αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την παροχή πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Ταμείου Προσαρμογής και τα μέτρα για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνουμε τη λειτουργία του Ταμείου Προσαρμογής και έχουμε πιο αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων του Ταμείου αυτού στο μέλλον. Χαιρετίζω επίσης και την διεύρυνση της εμβέλειας του Ταμείου αυτού σε σχέση με τους επιλέξιμους δικαίουχους, αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι αυτοαπασχολούμενοι και την παροχή υπηρεσιών που δίδονται από το Ταμείο προσαρμογή για άτομα τα οποία δεν είναι εργασόμενοι ή σε μαθητεία. Όταν ε, κάτω της ηλικία των 25 ή 30 υπό τη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Και επίσης για την ε, βελτίωση των πόρων που είναι διαθέσιμοι. Υποστηρίζω επίσης το να δοθεί περαιτέρω βοήθεια σε τοπικό επίπεδο για να δοθούν τοπικές λύσεις σε αντιμετώπιση καταστάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ταμείου προσαρμογή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το πετύχουμε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, γιατί αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο στην Ιρλανδία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην τοπική και περιφερειακή συμμετοχή των εμπλεκομένων. Θέλουμε επίση να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια στα κριτήρια του Ταμείου για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ε, ε, υποβολή αιτήσεων από περιοχέ και κομιτείε που έχουν χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού. Αλλά τονίζω ότι είναι ιδιαίτερο και εξαιρετικό ο χαρακτήρας αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει και ένα αιτήσιο κονδύλιο. Οι 500 εργασόμενοι ως κατόφλοι θα πρέπει να μειωθούν σε 200 για να μπορέσει να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στην υποστήριξη του Ταμείου αυτού. Και θέλω να υποστηρίξω επίσης την ανάγκη να επανέλθουμε τουλάχιστον στο προηγούμενο επίπεδο κονδυλίων του Ταμείου Προσαρμογής για 500 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει διευρυνθεί το, η σφαίρα εφαρμογής του ταμείου αυτού. Τέλος, με την αρχή της ενότητας του προπολογισμού πιστεύω ότι για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας είναι υψής της σημασίας να υποστηρίξουμε την ενσωμάτωση του Ταμείου Προσαρμογής στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση. Θέλω να τονίσω επίσης ότι είναι απαραίτητο να επανενσωματώσουμε το κριτήριο της εξαίρεσης κρίσης και να έχουμε ειδικά κονδύλια για την απελευθέρωση των κονδυλίων του Ταμείου αυτού στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σημαντικές δημοσιονομικές δυσκολίες και εδώ φυσικά μιλώ για χώρες όπως είναι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση και βρισκόνται ακόμα σε φάση λιτότητας. Η ανεργία και η απώλεια θέσεων είναι σε ιστορικό ρεκόρ, επίπεδο ρεκόρ στην Ιρλανδία και πολλά από τα μέρη της χώρας μας δεν έχουν πια νέους οι οποίοι υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν. Αυτό λοιπόν θα έχει μεγάλα προβλήματα για το μέλλον και τη βιωσιμότητα των πόλεων και των χωριών μας. Αυτό είναι λοιπόν ένα κατεπήγον πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και θα ήθελα να προτείνω η ενίσχυση όλων αυτών των ε, ε αιτήσεων να ληφθούν υπόψη και με εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για να υπάρξει η απαραίτητη υποστήριξη για τους εργαζόμενους και να υπάρχουν οι απαραίτητες πρόνοιες ώστε να μην υπάρχουν καταχρηστικές ε, εφαρμογές του Ταμείου αυτού. Το νομικό τώρα πλαίσιο και παρεχόμαστε σε αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές προηγουμένως σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και τη λογοδεσία. Το νομικό πλαίσιο έχει τροποποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2013, αλλά έκτοτε δεν έχουμε καμία αξιολόγηση για την ε, επίπτωση αυτής της αλλαγής και θα ήθελα να έχω κάποια αποτελέσματα σε επίπεδο αξιολόγησης και χαίρομαι για τις αλλαγές που έχουν αυξήσει την ε, εμβέλεια του προγράμματος αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Ο κύριος Μακά τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Είναι ανάγκη πράγματι να έχουμε μία εκστρατεία όσον αφορά το Ταμείο αυτό προσαρμογής στις ε, επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι χώρες ε, μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει συνειδητοποίηση, να μάθει ο κόσμος για το Ταμείο αυτό, γιατί οι χώρες μέλη μόνο να αποφεληθούν έχουν. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αναλάβει κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες και να χρησιμοποιηθούν και κονδύλια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, κυρίως για τους δικαιούχους και είναι πολύ καλό το ότι, έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πολύ γρήγορα δίνεται η βοήθεια αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, κυρία Οντή. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Όντω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το θέμα αυτό, τότε, δηλαδή οι περιφέρειες μπορούν να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση. Είναι μια προσθεθέμενη αξία στο κάτω-κάτω της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ότι τα χρήματα δηλαδή πηγαίνουν κατευθείαν σε αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται και εντοπίζονται έτσι πολύ καλύτερα οι πραγματικές ανάγκες που καλύπτονται. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο από ό,τι βλέπω. Οπότε θα περάσουμε τώρα στην τρίτη ανακοίνωση. Πρόκειται για την κινητοποίηση στη Ρουμανία. του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Κοσμιοποίηση με εισηγητή τον κύριο Μουσά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση αυτή αναφέρεται στην κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μετά από αίτημα των αρχών τη Ρουμανίας το Δεκέμβριο του 2012 για μια χαλιβουργία που ονομάζεται Κοντ Μέχελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο φέτος αποφάσισε ότι οι προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση αυτή καλύπτονται. Το λέω και στο σχέδιο εκθεσής μου ότι και εγώ συμφωνώ πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση αυτή. Όπως λοιπόν σας είπα, πρόκειται για μια χαλιβουργία και όπως γνωρίζουμε υπήρξαν ε, τεράστιες διαρθρωτικές αλλαγές στη Χαλιβουργία τα τελευταία χρόνια. Εν μέρη αυτό οφείλεται και στην οικονομική κρίση. Ή Ιδιαίτερα το για τα μεταπημένα ή για τα τελικά προϊόντα χαλιβουργίας, ο κλάδος αυτός επλήγει πάρα πολύ λόγω της κρίσης, γιατί οι Ευρωπαίοι παραγωγοί μειώθηκαν πάρα πολύ σε σχέση με τους αντίστοιχους στην Κίνα. Οπότε, πολύ συγκεκριμένα για την εταιρεία αυτή έπρεπε να απολύσει πάνω από 800 στη περίοδο αναφοράς Ιούνιο με Οκτώβριο δηλαδή του 2012 και πάνω από 600 νωρίτερα και μετά από την περίοδο αυτή αναφοράς. Πάνω από 1500 δηλαδή έχασαν τη δουλειά τους. Πάνω από χίλιοι μπορούν να αποφεληθούν από μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης, των, αναγκών μάλλον, είναι 700 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής. Ο στόχος είναι βέβαια να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ατόμων που απολύθηκαν, 1500 όπως σας είπα, με κατάρτιση, με επιμόρφωση, με βοήθεια οικονομική προκειμένου να ξεκινήσουν μια ατομική επιχείρηση, ή συνεταιρισμούς όπου να μπορούν να απασχοληθούν 250 το πολύ. Η δημιουργία μιας τέτοιας επιχείρησης πήρε βέβαια περισσότερο χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται και για μια καινοτομία η χρηματοδότηση αυτή από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δυόμιση χρόνια χρειάστηκε επίση η αξιολογήση του προγράμματο αυτού. Οι Ρωμανικέ Αρχέ πάντω το Δεκέμβριο του 2012 επέβαλαν το πρόγραμμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φω τον Μάιο του 2014. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι έμειναν στην ανεργία δύο χρόνια περίπου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς ως Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε γρήγορα. Όπως το είπατε και εσείς ε, πρόεδρε για την προηγούμενη έκθεση, οι προθεσμίες από πλευράς του Κοινοβουλίου ισχύουν και για την έκθεση αυτή. Οπότε 4 Σεπτεμβρίου προθεσμία για υποβολή τροπολογιών και η απόφαση στην Επιτροπή μας 11 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε τη βδομάδα 15-16 Σεπτεμβρίου, τη βδομάδα εκείνη. Λοιπόν, με δύο λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε θετική σύσταση, το συμπεριλαμβάνω και εγώ στην εκθεσή μου. Τα ωφέλη, όπως σας είπα, αφορούν χίλιους εργαζόμενους, είναι πάρα πολύ συγκεντρημένα τα ωφέλη αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί επλήγησαν εξαιτία της ε, κρίσης και της παγκοσμιοποίησης. Ένα τελευταίο πράγμα. Το 1 τρίτο του εργατικού δυναμικού στην περιφέρεια αυτή εξαρτόταν από την χαλιβουργία αυτή, τη συγκεκριμένη δηλαδή επιχείρηση, το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Πάντω οι υπηρεσίε απασχόληση, οι τοπικέ στη Ρουμανία πρέπει να ξέρετε ότι έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν προγράμματα όπω αυτά τα οποία σα ανέφερα πριν. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Μούρσαν. Οι απολύσει έγιναν το 2012. Ναι, το 2012. Ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε πως πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία παραπάνω, γιατί μένουν πολύ καιρό οι άνθρωποι στην ανεργία έτσι. Δύσκολα παίρνει πάλι μπρος η μηχανή. Ο κύριος Ντελανό έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την έκθεση αυτή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές οι αλλαγές που γίνονται τελευταία και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, όχι μόνο Χαλιβουργία, τη Ρουμανία τη γνωρίζω, όπως και άλλες χώρες, γνωρίζω τις περιπτώσεις αυτές πολύ καλά. Είμαστε σε μια περίοδο λοιπόν αλλαγών όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Συνεπώς πρέπει να συνοδεύσουμε τον κόσμο, να στηρίξουμε τον κόσμο που πλήττεται από τις αλλαγές αυτές. Αλλά πρέπει να δουλεύουμε και θετικά υπέρ ε, της δημιουργίας νέων υλικών. Εντάξει, όχι δικιά μας η Επιτροπή, αλλά εδώ και πολύ καιρό εγώ μιλάω για αυτό το θέμα. Σήμερα υπάρχουν είτε είναι κεραμικά, είτε με άνθρακα υλικά, τα οποία θα έχουν πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά από αυτά που έχει ο Χάλιβας μέχρι τώρα και που θα αλλάξουν παντελώς το βιομηχανικό τοπίο της Ευρώπης. Πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Εδώ είναι εμβληματική η έκθεση αυτή εξαιτία ακριβώς των αλλαγών που υφίσταται η Ευρώπη. Κύριος Νεγρέσκου. Καλημέρα συμφωνώ και εγώ με την πρόταση για τα κονδύλια αυτά. Θέλω όμως να σας προσθέσω κάποια στοιχεία εδώ. Εγώ έρχομαι από την Τρασιλβανία, εκεί δηλαδή που υπήρχε αυτό το εργοστάσιο. Θα ήθελα η έκθεση να αναφέρει ότι πρόκειται για 17 μήνες από τότε που υπευλήθη το αίτημα από τις ρουμανικές αρχές είναι πολύ μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα να το συγκρίνουμε με τις άλλες περιπτώσεις. Οι άλλες περιπτώσεις, οι αιτήσει υποβλήθηκαν το 2014. Ενώ εδώ πέρα έχουμε και τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που επλήγησαν και άρα χρειάζονται τη βοήθεια, αλλά πρόκειται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να ληφθεί η θετική απόφαση. Και κάτι ακόμα που πρέπει να πάρουμε υπόψη και πρέπει να βάλετε στην έκθεσή σας, πιστεύω, ότι χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πότε ακριβώς θα δοθούν τα χρήματα. Ήδη έχουν περάσει 17 μήνες. Ας βάλουμε και μια ημερομηνία λοιπόν στην έκθεση αυτή. Και μια που μιλάμε για τόσο μεγάλη καθυστέρηση, θα έπρεπε την κατάσταση τότε με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Στους 17 αυτούς μήνες άλλαξαν κάποια πράγματα, πληθωρισμός, μειώθηκε αγοραστική δύναμη κλπ. Το ποσό αυτό δηλαδή πρέπει να διορθωθεί για να λάβει υπόψη και τους παράγοντες αυτούς, τις αλλαγές αυτές. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η Μέκελ ήταν μια ρωσική εταιρεία. Πολύ συχνά θα δούμε πολλές ρωσικές επιχειρήσεις να κλείνουν οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι έτσι καταλήγουν στην ανεργία. Εμείς που είμαστε ευρωβουλευτές πρέπει να προσέξουμε το φαινόμενο αυτό, το οποίο θα συναντάμε όλο και πιο συχνά, και να συμπεριλάβουμε και την πραγματικότητα αυτή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ταφαντέρ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ έρχομαι από τη Ρουμανία και όπως ξέρετε αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Εδώ και 17 μήνες είχε ζητήσει τα κονδύλια αυτά η Ρουμανία και ζήτησα από τον εισηγητή στην έκθεση του να τονίσει την ανάγκη να εκταμιευτούν αυτά τα ποσά τα ταχύτερο να το μιλάμε για χίλια άτομα όπως λέει επίση η έκθεση μιλάμε για μια περιοχή που έχει μονάχα μία οικονομική δραστηριότητα. Δεν είναι μονάχα τα, 15, τα 1500 άτομα τα οποία έμειναν άνεργα. Μιλάμε για 1500 οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει την πηγή εισοδήματός τους. Δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες απασχόλησης στην περιοχή αυτή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορεί να κάνει κανείς. Σας ζητώ λοιπόν να υποστηρίξετε αυτή την έκθεση και ας προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα μπορούσαμε με τον τρόπο αυτό να δώσουμε και ένα θετικό παράδειγμα και υπογραμμίζω και πάλι ότι έχουν περάσει 17 μήνες χωρίς να υπάρξει συνέχεια στην αίτηση αυτή. Ας επιταχύνουμε τη διαδικασία. Είναι σημαντικό για τη Ρουμανία αλλά και για όλη την Ευρώπη να υπάρξει μια λύση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μανκά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι φανερό ότι θα υποστηρίξω και εγώ αυτό το μέτρο. Είναι μια πάρα πολύ τυπική αίτηση για βοήθεια, αλλά έχει και καινοτόμα χαρακτήρα. Θα μπορέσουν να επωφεληθούν οι εργαζόμενοι από τη χρήση νέων μορφών εξοπλισμού και τεχνολογίας και αυτό θα βοηθήσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι πολύ θετικό αυτό. Μπορούμε ενδεχομένως να κάνουμε και μια αξιολόγηση μετά από παρέλευση δύο ετών. Νομίζω ότι θα εκμεταλλευτούν πολύ θετικά αυτή τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι εφόσον του δοθεί. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Θέλετε να υπάρξει μια αξιολόγηση των δαπανών και των πληρωμών που θα δοθούν. Μπορούμε να περάσουμε στην τέταρτη αίτηση για την εφαρμογή του Ταμείου αυτού 2014-003 Αραγωνία, Τρόφιμο και Ποτά στην Ισπανία με ε, εισηγήτρια, την κυρία Γιάχτεμακή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω φιλανδικά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ισπανία έκανε μια αίτηση το Φεβρουάριο για τη χρηματοδότηση αυτή και όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές θέλω να τονίσω ότι θα μπορούσε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Έχουν περάσει ήδη 17 μήνες από τότε που κατατέθηκε αυτή η αίτηση. Και μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ληφθεί κατά πάσα μια απόφαση, θα έχουμε φτάσει στους 24 μήνες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η Ευρώπη μπορεί να θεωρήσει ότι προχωρεί με γρήγορου ρυθμού. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Η αίτηση αυτή έχει να κάνει με την περιοχή της Αραγωνίας στην Ισπανία, όπου ο τρομέα των τροφίμων και ποτών στην περιοχή αυτή έχει πληγεί ιδιαίτερα λόγω της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης που ήταν ιδιαίτερα σοβαρή κρίση και σε αυτή την περιοχή. Μιλάμε για 204 ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει άνεργοι. Πρόκειται για μια αίτηση που έχει να κάνει με την επανεκπαίδευση ατόμων από αυτή την περιοχή. δεν ξέρω τι έχει γίνει ενδιαμέσως, γιατί βέβαια έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ξέρουμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει μια ανθρώπινη τραγωδία το γεγονός ότι δεν ανέλαβε κανείς δράση για τα θέματα αυτά. Χρειάζονται 960.000 ευρώ και 60% του συνολικού κόστους θα πάει για να καλύψει τις ανάγκες των ανέργων. Υπήρξαν δύο αιτήσει το 2010 και το 2012 όπου υπήρχαν προβλήματα με την διάρθρωση του τομέα και την κρίση στην λιανική αγορά τροφίμων και ποτών. Η ανεργία στην περιοχή αυτή έχει φτάσει από 14% στο 19% πρόσφατα, σύμφωνα με τις ε, στατιστικές της Κομισιόν, σύμφωνα με την ε, έκθεση της Κομισιόν εκπληρεί όλα τα απαιτούμενα η περιοχή της Αραγωνίας και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως. Αλλά και η διαδικασία είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί για αυτήν την περίπτωση, ιδίως άμα σκεφτούμε ότι ο στόχος εδώ είναι να προωθήσουμε την επανεκπαίδευση ανέργων και τα συνοδευτικά μέτρα που θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά να έχουν μια θέση εργασίας είτε στην περιοχή αυτή είτε κάπου αλλού Επομένως έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα μόνο αυτής της ε, ε, αίτηση αλλά και άλλων αιτήσεων και πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ετσιανίκουε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, σε σχέση με αυτή την αίτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, θα ήθελα να πω το εξή. Και εγώ έρχομαι από την Αραγωνία συγκεκριμένα. Έχω δει στην ίδια μου την πόλη πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα αυτό με, ε, με μαγαζιά και μικρές επιχειρήσεις να κλείνουν. Γνωρίζω πολύ καλά προσωπικά πολλά άτομα τα οποία εργαζόντουσαν στον τομέα αυτό και εργαζόντουσαν στον τομέα το, της ε, εστίασης και των ε, ξενοδοχείων που έχουν περάσει πολύ δύσκολες ε, στιγμές που δεν θέλω να τις περάσει κανένα άλλο άτομο στον κόσμο και γι' αυτό θέλω να τονίσω την ανάγκη να κινητοποιηθούν το ταχύτερο αυτά τα κονδύλια και να εγκριθεί αυτή η αίτηση. Επίσης όμως θα ήθελα να αναφέρω ότι διάβασα όλο το σύνολο όλο τον κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από τα μέτρα αυτά και γνωρίζω από πρώτο χέρι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν είναι λοιπόν κάτι το τυχαίο αυτό, αλλά μου δίνει μια πολύ καλή εικόνα για την έκταση αυτού του προβλήματος το οποίο σοβεί τώρα στην Ισπανία και φυσικά πιστεύω το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες χώρες του Νότου της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να τονίσω ότι πρέπει να δώσουμε τη βοήθεια στα άτομα αυτά τα οποία περνάνε πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και γενικότερα για τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης και της ε, ε κρίσης αυτής που είναι σαν μια φυσική καταστροφή και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Δεν πρέπει όμως να την αντιμετωπίσουμε μόνο όταν συμβαίνει αυτή η τραγωδία, πρέπει ως ευφυή άτομα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την πρόληψη τέτοιων κρίσεων και τέτοιων καταστροφών στο μέλλον. Και αυτό φυσικά συνδέεται με κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε που είναι η Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου με τις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Κενίκουε. Είναι αλήθεια ότι θα ήταν ε, πιο φρόνιμο να προβλέψουμε τις ε, προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να προετοιμαστούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές και όχι να παρεμβαίνουμε ε, κατόπιν εορτής όπως τώρα. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητά το λόγο για όσον, όσον αφορά την Ραγόν, όχι. Περνάμε λοιπόν στην πέμπτη ε, ανακοίνωση για το EGF ε, e πάλι 002-2014 ε, για την Ολλανδία Gelderland over Eisel. Πεντών. Ευχαριστώ. Είμαι καινούριο εδώ στο Κοινοβούλιο. Και με εκπλήσει ήδη το πόσα χρήματα ήδη δίνονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Εξέτασα αυτή την περίπτωση και διαπίστωσα ότι καλώς δαπανήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Ολλανδία βλέπετε όπω πολλέ άλλε χώρε επλήγει και εκείνη από την οικονομική κρίση. Ιδιαίτερα ο κατασκευαστικό τομέα, κατασκευή κτηρίων μάλιστα. Ε, δεν χτίζονται πια καινούργια σπίτια, κυρίως γιατί οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν ενυπόθηκα δάνεια πια. Αυτό σημαίνει ότι και οι τιμές των σπιτιών έχουν πέσει πάρα πολύ, αλλά δεν κατασκευάζονται και νέα σπίτια. Ο οικοδομικό τομέας λοιπόν επλήγει πάρα πολύ σοβαρά στην Ολλανδία. Είναι επίσης αλήθεια ότι και στην περιφέρεια της χώρας υπάρχουν ε, ε, προβλήματα. Διαφορά υπάρχει βέβαια ανάμεσα στο κέντρο της χώρας και την περιφέρεια. Στο κέντρο της χώρας κάτι γίνεται, κάποια ανάκαμψη αρχίζει να εμφανίζεται, αλλά στην περιφέρεια όχι. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτό που τώρα μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη ανεργία, μπορεί κάλλιστα να καταλήξει σε μακροχρόνια ανεργία. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην κατασκευή κτηρίων όπου υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις με αυτοπασχολούμενους, άνθρωποι οι δεν έχουν ιδιαίτερα προσόντα, δεν έχουν μεγάλη μόρφωση. Αυτοί λοιπόν είναι που χρειάζονται πραγματικά στήριξη για να μπορέσουν να ξαναβρούν δουλειά στην Ολλανδική αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν είναι καλά στοχευμένη η πρόταση αυτή στην περιφέρεια της χώρας και φαίνεται να είναι κάτι πολύ αποτελεσματικό γιατί τα χρήματα πράγματι πηγαίνουν για να βρει ο κόσμος δουλειά ώστε οι άνεργοι να μπορέσουν να ξαναβρούν δουλειά στην Ολλανδική Αγορά Εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλή πρόταση και συμφωνούμε απόλυτα με αυτήν. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγήτα. Και τώρα για να καλέσω όσους θέλουν να το σχολιάσουν να το κάνουν τώρα. Δεν ζητά κανείς το λόγο. Οπότε περνάμε στις πληροφορίε που είχαν προβλεφθεί. Α, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και για τι τέσσερι αυτέ εκθέσει όπου ακούσαμε για το πρόβλημα τις ε, καθυστερημένες δράσεις όσον αφορά τη χορήγηση αυτών των κονδυλίων στα κρατήματα. Θα ήθελα να προτείνω λοιπόν να βρούμε τους λόγους τους οποίους οφείλεται αυτή η καθυστερημένη δράση και επίσης να διερευνήσουμε λύσεις για αυτές, να, να, να εξελιχθούν αυτές οι καθυστερήσεις. Θα ήθελα να πω ότι οι συγητές εδώ, ε, αλλά και οι μελλοντικοί συγητές για αυτές τις, ε, αυτού του είδους τις εκθέσεις, όταν θα προκύπτουν προβλήματα με το Ταμείο και την κόρηση ε, των κονδυλίων να περιλαμβάνουν στις εκθέσεις τους τις συνέπειες ε, αυτής της αργής ε, διεκπαιρέωσης αυτών των αιτήσεων. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε μήπως λόγω της παγκοσμιοποίησης τέτοια προβλήματα εξακολουθήσουν να προκύπτουν και να διαρωτηθούμε λοιπόν κατά πόσο το Ταμείο έχει αρκετά κονδύλια στη διάθεσή του ώστε να μπορέσει να ε, αντιμετωπίσει αυτές τις ε, επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης αλλά με ταχύτερο ρυθμό. Ευχαριστώ. Ναι, είναι αλήθεια ότι καθένας από τους εισηγητές ε, διατύπωσε επικρίσεις, ότι υπάρχει ένα είδος αδράνεια σε μια υπερβολική απόσταση ανάμεσα στις οδυνηρές αυτές καταστάσεις που ε, καλούν ε, τη κινητοποίηση του Ταμείου για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης, ε, την, την κατάρτιση του φακέλου, τις ψηφοφορίες που πρέπει να γίνουν και ανησυχούμε για τις πληρωμές και την καταβολή αυτών, γιατί και εκεί ξέρουμε πόση καθυστέρηση υπάρχει. Οπότε, απέναντι σε αυτή τη χιονοστιβάδα επικρίσεων λοιπόν, ίσως θα πρέπει η Κομισιόν να μας πει τα σχόλιά της, τις παρατηρήσεις της, για να μας καθησυχάσει ίσως. Κυρία Γενική Διευθύντρια. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Όντως, σκόπευα να μην πάρω το λόγο, αλλά επειδή τόσοι πολλοί βουλευτές μίλησαν για το θέμα των καθυστερήσεων, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τρία ζητήματα. Καταρχήν, να πω ότι, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν νέοι κανόνες που ισχύουν και μειώνουν το χρόνο για τη λήψη αποφάσεων σε αυτού του είδους τα αιτήματα. Στην περίπτωση νέων αιτήσεων η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέσα σε μια περίοδο τεσσάρων μηνών. Η πρώτη υπόθεση στην οποία αναφερθήκαμε, η ρουμανική περίοδο, ενέπιπτε στους παλιούς κανόνες ε, που προέβλεπαν μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε εκείνη την περίπτωση και ο ίδιος ο εισηγητής νομίζω αναγνώρισε πως η δυσκολία συνδυόταν με τη δημιουργία του συνεταιρισμού. Έπρεπε να επαληθεύσουμε ότι όντως πρόκειται για ένα βιώσιμο ε, σχέδιο, ότι θα υπήρχε ζήτηση για αυτά τα και ότι ο κόσμος πραγματικά θα συμμετείχε στο συνεταιρισμό. Αυτό είναι η βασική εξήγηση για την καθυστέρηση στη συγκεκριμένη ε, περίπτωση. Δεύτερη μου παρατήρηση για την Ισπανία τώρα. Ίσως να υπήρξε κάποια παρεξήγηση, διότι η αίτηση αυτή έγινε σε Φεβρουάριο του 2014. Δεν είναι και τόσο μεγάλη καθυστέρηση αυτή την υπόθεση. Το τρίτο μου σχόλιο είναι ότι από τη στιγμή που οι δύο δημοσιονομικές αρχές συμφωνήσουν, τότε περνάνε δύο εβδομάδες ώστε η Κομισιόν να καταβάλει τα ποσά. Ε, μπορώ, λοιπόν, δεν μπορώ παρά να στηρίξω τις παρατηρήσεις του Προέδρου να προσπαθήσει να ληφθεί η απόφαση στο Κοινοβούλιο όσο γίνεται πιο σύντομα, ώστε να εκτελεστούν αυτέ οι αποφάσει όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το μπαλάκι είναι στο δικό μας γήπεδο, το κοινοβουλίο. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπο κατάρτισης των αιτήσεων και ψηφοφορίες πιο γρήγορα γιατί όταν μένεται η φωτιά δεν ε, ρωτάμε το Δημοτικό Συμβούλιο αν πρέπει να, πάνε, να στείλει πυροσβέστες. Σε αυτές τις ε, έκτακτες και τόσο δυνηρές λοιπόν καταστάσεις θα πρέπει να βρούμε τρόπο να επιταχύνουμε τη διαδικασία λήψης απόφασης και καταβολής των, δαπάνω, των πληρωμών αυτών. Μάλιστα, ωραία, ολοκληρώσαμε αυτές τις πέντε αιτήσει ε, κινητοποίησης του Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και Φτάνουμε στις ψηφοφορίες. Οι εισηγητές είναι ο Ζηράς Δεπρέ και η κυρία Χολμάγερ. Να τους συμβουλευτών για να ρωτήσω αν μπορούμε τώρα να περάσουμε στην εξέταση των ανακοινώσεων και στις ψηφοφορίες, διότι η ψηφοφορία είχε προβλεφθεί για τις 12 και 10 και ίσως ορισμένοι από τους συναδέλφους μας να έχουν προβλέψει να φτάσουν στις 12 και 10. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες αυτές. Κύριε Ντεπρέ, εσείς τι λέτε. Κύριε Πρόεδρε, έχω σκοπό να προχωρήσουμε γρήγορα. Ναι, εγώ νομίζω πως μπορούμε να ψηφίσουμε εδώ, αν δεν υπάρχει αντίρρηση από πλευρά των συναδέλφων, στις 12 και 10 ή στις 12 και 10. 12 και 10 ή 12 και 12 εάν δεν έχετε αντιρρήσεις να τις ψηφίσουμε πολύ γρήγορα. Από μένα πάντως δεν υπάρχει αντίρρηση. Κύριε Χολμάγερ, έχετε εσείς αντίρρηση? Όχι. Ναι, 10 λεπτά να γεμίσουμε το χρόνο, αυτό είναι. Ναι, ναι. Μια πάρα πολύ σύντομη επεξήγηση είναι για το, την αρχή προστασία των προσωπικών δεδομένων. Χρειάζεται μία μεταφορά πιστώσεων. Μία θέση η οποία θα μετατραπεί από θέση ε, προσωρινού υπαλλήλου, μάλλον με σύμβαση σε μία θέση κανονικού υπαλλήλου. Αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα λοιπόν. Δεύτερον, έχουμε μια αίτηση από την Επιτροπή Περιφερειών ένα προ... μια τροποποίηση θέσης προσωπικού για, την... Ε, για τον παιδικό σταθμό. Είναι η φυσιολογική διαδικασία στην Επιτροπή των Περιφερειών για να μπορούν τα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής των Περιφερειών να πηγαίνουν στον παιδικό, να στέλνουν τα παιδιά στον παιδικό σταθμό άλλο θεσμικό οργάνο και να μεταφέρουν λοιπόν χρήματα προς την κατεύθυνση αυτή και η τρίτη μεταφορά αφορά πάλι την Επιτροπή των Περιφερειών και πρόκειται για μια τροποποίηση στο οργανόγραμμα. Είναι μια απόφαση η οποία έχει ήδη ληφθεί. για ένα ε, μέλος του προσωπικού που έχει μεταφερθεί σε μια πολιτική ομάδα και επομένως η θέση του θα πρέπει να καλυφθεί. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία ζήτησε η Επιτροπή των Περιφερειών. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος, ο Ζωάν Πρέ. Πάρα πολύ σύντομα κύριε πρόεδρε, έχουμε πάρει ένα μεγάλο πακέτο προτάσεων μεταφορών. Κάποιες από αυτές τις μεταφορές μπορούν να ψηφιστούν αργότερα. Είναι οι προτάσεις 12, 13, 14, 15 και 16. Αυτές λοιπόν θα αντιμετωπιστούν στην επόμενη μας συνεδρία. Θα σας παρουσιάσω τις προτάσεις που μπορούν να ψηφιστούν σήμερα. Καταρχήν τη μεταφορά πιστώσεων υπαριθμών 11 που αφορά μια επαλεξισορρόψη για το 2014 διοικητικών δαπανών για τους αποκεντρωμένους φορείς. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ρυθμίσει η Κομισιόν. Υπάρχει μετά η μεταφορά 18, πρόκειται για μία προκαταβολή η οποία θα ε, επιστραφεί το 2015 για μία ε, υποστήριξη προς το Συμβούλιο ε, για την εξυγίανση των τραπεζών που θα λειτουργήσει από το 2015. Από το 2015 θα χρηματοδοτείται από συνεισφορές των, τραπεζών και θα επιστραφεί η προκαταβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά έχουμε τη μεταφορά 19. Έχουμε την νομική βάση για το πρόγραμμα Horizon 2020 που τροποποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2013 μετά από την έγκριση του προπολισμού του 2014 πρέπει να τροποποιηθούν οι πιστώσεις υποχρέωσης για να ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις που ελήφθησαν το Δεκέμβριο του 2013 σε σχέση με τη νομική βάση. 20.000 2014. Είναι μια <clears throat> μεταφορά που θα επιτρέψει στη Σερβία και το Μαυροβούνιο να κάνουν την καλύτερη χρήση των πιστώσεων υποχρεώσεων που είναι διαθέσιμα στο εργαλείο προενταξιακής ε, ε, βοήθειας για να βελτιωθεί καλύτερα η χρηματοδότηση των προγραμματών αυτών. 21-2014, και αυτό είναι προβληματικό, είναι μια μεταφορά 50 εκατομμύριων ευρώ από το αποθεματικό και την ε, ε, έκτακτη βοήθεια στο ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Συρία. 22-14, 125 εκατομμύρια σε πιστώσεις υποχρέωσεων και 7 σε πιστώσεις πληρωμών για τη Συρία και οι γειτονικέ χώρες για να βοηθήσουμε την αντιμετώπιση της ροής των προσφύγων στη Συρία και σε γειτονικέ χώρες. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε είναι 12 και 7 όπως καταλάβατε. Σας ευχαριστώ και τους δύο σας για τις διευκρινήσεις. Υπάρχουν σχόλια σε σχέση με τα θέματα αυτά. Έχουμε πέντε λεπτά για να κάνουμε τα σχολιά μας, εάν θέλετε. Εάν όμως δεν υπάρχουν σχόλια, μήπως θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε. Να επιταχύνουμε τη διαδικασία, αν δεν βλέπετε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ίσως μπορούμε, εφόσον έχουμε καταγγείλει την αδράνεια του συστήματος, να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού όλες τις, τις αποφάσεις 11, 18, 19, 20, 21 και 22 που παρουσίασε ο κ. Ντεπρέμ. υπέρ υπέρ διανατάσεις χειρών ευχαριστώ κατά δεν υπάρχουν αντίθετες θέσεις αποχές μία μία δύο αποχές ευχαριστώ ούτως απεφασίστε λοιπόν τα άλλα τμήματα του προπολογισμού που παρουσιάστηκαν από την κυρία Χολμάια για την Επιτροπή Περιφερειών. Τη μεταφορά 1-2014. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Απεφασίστη για τον επόπτη προσωπικών δεδομένων η μεταφορά EDPS παριθμών 1 υπέρ ευχαριστώ κατά αποχές δύο αποχές και τέλος τελευταία απόφαση την Επιτροπή των Περιφερειών τροποποίηση του οργανογράμματος 2014 υπέρ κατά όχι αποχές δύο αποχές έχουμε κλείσει λοιπόν με την ημερησία διάταξη έχετε να θέσετε άλλα ερωτήματα όχι θα διακόψουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας και επανερχόμαστε στις 3 για να ακούσουμε την τρόικα των αποκεντρωμένων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λήξη της συνεδρίας. Θα τα πούμε.